Καλημέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Καθίστε παρακαλώ. Y guarden silencio, por favor. Καθίστε και λίγη ησυχία παρακαλώ. Continuamos con el orden del día. El punto número 10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 Τροπολογία 1 του εισηγητού, άρχεται ψηφοφορία, σύνδεση υπερπόντιων χωρών και ταφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά, το κάνουμε διανατάσσεως της χειρός. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ διανατάσσεως της χειρός. Κατά. Κανένας κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η πρώτη τροπολογία και μοναδική. Ψηφίζουμε το σύνολο της ονομαδότητας. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, μία αποχή. Εγκρίνεται και συγχαρητήρια στο συντάκτη της γνωμοδότης, τον κύριο Ριβελίνη. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο, το 11. Αλληλευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται Συμφωνία Αλληλευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης. Θα θυμάστε ότι πέρυσι το Μάιο ε, το νέο πρωτόκολλο για μια διετία. Το Νοέμβριο έγινε η παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα τέλη Νοεμβρίου έγινε η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό. Και σήμερα θα εξετάσουμε το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Ριβελίνη, στον οποίο δίνω και το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη συνοψίσατε το θέμα αυτό της συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαδαγασκάρης για την Αλία που επισέρχεται σειρά συμφωνιών που έχουν συναυθεί με τις χώρες του Ινδικού ωκεανού για την αλία του τόνου. Το πρωτόκολλο καθορίζει τη δυνατότητα αλίας για τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και καθορίζει την οικονομική αντιστάθμιση ε, που έλυγε το τέλος 2012. Οπότε χρειάζεται ένα νέο πρωτόκολλο όσον αφορά τις ε, απαιτήσει για τους στόλους μας. Η συμφωνία της εταιρικής σχέσεως εφαρμόζεται για μια διετή περίοδο, 2013-2014 και προβλέπει τη δυνατότητα αλίας για 96 σκάφη. 40 σκάφη αλήφθη τόνη και 26 αλευτικά σκάφη με ε, παραγάδι. Και αντιστάθμιση οικονομική που είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο με αύξηση 328.000 ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία. Εκεί συμπεριλαμβάνονται 975.000 ευρώ για την πρόσβαση στην ζώνη αλίας της Μαδαγασκάρης που αντιστοιχεί τα αφορά 15.000 τόνων το χρόνο, μια αύξηση 1.700 τόνων το χρόνο σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία και 550.000 ευρώ για ανάπτυξη ε, πολιτική ε, αλληλευτικής ε, από πλευρά τη Δημοκρατία Μαδαγασχάρης. Συνοψίζοντα, λοιπόν η αύξηση ποσοτική τη ποιότητα αναφορά συνδέεται και μια αύξηση τη οικονομική χρηματική αντιπαροχή και εξάλλου η αύξηση των αλλιευμάτων πραγματοποιείται σε απόλυτη συμφωνία με τι εγκυρότερε επιστημονικέ νομοδοτήσει τη Επιτροπή Διαχείριση τη Τόνους Τόνου του Ινδικού Ωκεανού. Εν τούτης, όσον αφορά τη χρησιμοποίηση στο πλαίσιο της παρούσης συμφωνίας αλληλευτικής σύμπραξης των οικονομικών πόρων χρειάζεται να πραγματοποιηθούν εξωτερικοί οικονομικοί έλεγχοι, εξωτερική, εξωτερικά όντι, τόσο να εξετάζονται οι δηλούμενες ε, δαπάνες. Εξακριβώνται οι δαπάνες οι πραγματικές. Φτάνουμε στο κομβικό σημείο της συζητήσεως που είναι το θέμα της πολιτικής κατάστασης στη Μαδαγασκάρη, που παραμένει ε, τεταμένη, ακόμα και αν υπάρχει ένας οδικός χάρτης, χάρτης πορείας για τον τερματισμό της κρίσης στη Μαδαγασκάρη, και αυτός ο χάρτης πορείας προβλέπει τις επόμενες προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές που θα γίνουν Μάιο και Ιούλιο παρουσία παρατηρητών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχει συσταθεί ανεξάρτητη επιτροπή εκλογών. Πέρα αυτού, ο μεταβατικός πρόεδρος, ο σωήνος πρόεδρος ε, της Ματαξάρης που είναι στην εξουσία από το 2009 μετά από πραξικόπημα στατιωτικό που έγινε, ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες ότι δεν θα είναι υποψήφιος για τις επικείμενες προεδρικές εκλογές και αυτό χάρη στις διεθνείς πιέσεις ε, που ασκήθηκαν από 15 μέλη της κοινότητας ανάπτυξης ε, της ε, Βορειοαφρικής ε, είναι πολύ, ε, της Νοτιού συγγνώμη, είναι μια πάρα πολύ καλή προσέγγιση όσον αφορά την μετάβαση στην πολιτική. Ε, ήρθα σε επαφή και με άλλους για να ετοιμάσω αυτή τη γνωμοδότηση που ελπίζω ότι θα την αποδεχτείτε και λέμε ότι είναι σημαντικό από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω να αποσταλεί θετικό μήνυμα υποστήριξη προ την Μαδαγασκάρη ε, εγκρίνοντας αυτή τη νέα συμφωνία για τη σύμπραξη όσον αφορά την αλληλεία σε μια στιγμή που ε, εξαρτάται ο υπολογισμό της δημοκρατίας της Μαδαγασκάρης από την διεθνή βοήθεια. Ευχαριστώ. Ωραία. Ποιος θέλει το λόγο, κύριε Λόβιν. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Ριβελίνη για την παρουσίασή σας αυτή. Έξοχη έκθεση. Είμαι η συντάκτρια της γνωμοδοτήσεως στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Συζητήσαμε χτες αυτή την ε, συμφωνία στην Επιτροπή μας και έχω δύο προβλήματα όσον αφορά αυτή τη συμφωνία. Η μία ανησυχία μικρότερη από την άλλη. Καταρχά το θέμα τη ρήτρα εμπιστευτικότητα με απασχολεί. Είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που έχει εισαχθεί στη συμφωνία με τη Μοζαμβίκη και με τον Μαυρίκιο και στην παρούσα συμφωνία. Εκεί αναφέρεται στο άρθρο 11 ότι οποιαδήποτε στιγμή όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με το σκάφη τη Ευρωπαϊκή Ενώση και τι αριθμητικέ δραστηριότητε στα ύδατα τη Μαδαγασκάρη θα θεωρούνται ω εμπιστευτικά και θα αντιμετωπίζονται τέτοια. Αυτό είναι μια διατύπωση που πηγαίνει πολύ μακριά. Το συζητήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή χτε, την Επιτροπή Ανάπτυξη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξήγησε ότι επρόκειτο μόνο περί εμπορικών στοιχείων και όσα σχετίζονται με τον ανταγωνισμό μεταξύ διαφόρων στόλων. πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να διατυπωθεί ούτω ώστε να δηλώνει ακριβώς ε, αυτό που πρέπει να δηλώνει. Δηλαδή αναφέρεται στην πρόσπιση των εμπορικών στοιχείων και όχι όλων των στοιχείων που αφορούν τα σκάφη τη της Ευρωπαϊκής και τις αλληλευτικές δραστηριότητε. να διαβάσετε τη διατύπωση, ε, δεν δίνεται δυνατότητα ούτε στην κοινωνία των πολιτών να γνωρίζει πόσα σκάφη αλλιεύουν, πού αλλιεύουν και τι. Αυτά θα έπρεπε να είναι διαθέσιμα στον κοινό. Αυτό το, το μικρό μου πρόβλημα, το μεγάλο μου πρόβλημα τώρα. Αυτό αφορά το εξής η Μαδαγασκάρη μετά το πραξικόπημα του 2009 έχει αναστείλει την αναπτυξιακή συνεργασία του άρθρου 96 της Συμφωνίας Κοτονού. Καμία αναπτυξιακή βοήθεια δεν χορηγείται στη Μαδαγασκάρη διότι δεν έχει αποκατασταθεί η δημοκρατία, ο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτο δικαίου στη χώρα. Και αυτό ακριβώς αφορά ε, το άρθρο 96 τη Συμφωνία Κοτονού. Περί αυτού πρόκειται. Αναμένονται εκλογέ τον Μάιο. Υπέροχα. Και άκουσα και πολύ καλές ειδήσει. Δηλαδή ότι ο τωρινό πρόεδρος δεν θα είναι υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές, που και αυτό ήταν προπόθεση. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, Όμω υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητε όπως οι πολιτικοί εξόριστοι να μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα και να ψηφίσουν. Υπάρχουν εκκρεμότητε ακόμα. Το βασικό μου πρόβλημα για να δώσω συμφωνία στη συμφωνία πριν από τις εκλογές είναι το εξής. Είναι παράλογο να δώσουμε σύμφωνη γνώμη για μια συμφωνία με ένα πρωτόκολλο το οποίο αυτό καθε αυτό λέγει ότι θα έπρεπε να υπάρξει αναστολή του πρωτοκόλλου Σύμφωνα με το άρθρο 9 της Συμφωνίας Κοτονού ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 8 και 96 της εν λόγω συμφωνίας. Εν τη αυτή η περιπτώση όλα τα εθνικά σκάπη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και οι δραστηριότητε τους στα ύδατα της Μαδαγασκάρης θα ανασταλούν. Δηλαδή, ποια είναι η κατάσταση. Όλα έχουν ανασταλεί δυνάμει τη Συμφωνίας Κοτονού και μετά πρέπει να ψηφίσουμε ναι για ένα πρωτόκολλο που λέει ότι αν δεν υπάρξει ε, δημοκρατία πρέπει να ανασταλεί η Δεν ε, έχει νόημα αυτό καθόλου. Είναι εντελώς παράλογο. Ε, δεν μπορούμε να συνενέσουμε σε κάτι σύμφωνα όταν δεν υπάρχει βάση συμφωνία, μπορούμε να συμφωνήσουμε τη συμφωνία και να αναστείλουμε το επόμενο λεπτό. Δεν το βρίσκω καθόλου λογικό. Η Επιτροπή Ανάπτυξη πιστεύει, εγώ πιστεύω, να συνενέσουμε όσον αφορά τη συμφωνία, αλλά μετά τι εκλογέ, μετά τη διενέργεια των εκλογών. Τίποτα δεν μα υποχρεώνει να εγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία, δίποτε λευτική συμφωνία εντό συγκεκριμένη χρονική περίοδου. Ξέρετε τι έγινε με το Μαρόκο. Χρειαστήκαμε περίπου ένα χρόνο μετά την θέση ισχύ του πρωτοκόλου. Τότε ψήφισε το Κοινοβούλιο. Άρα δεν υπάρχει βιασύνη. Δεν πρέπει να βιαστεί να ψηφίσει το Κοινοβούλιο. Ο κύριος Κάσμαν της Σοσιαλιστικής Ομάδας στην Επιτροπή Ανάπτυξης ανησυχούσε πάρα πολύ διότι είναι εισηγητής για την Συμφωνία Κοτονού και πιστεύει ότι αν υπερψηφίσουμε αυτή τη συμφωνία όταν μια χώρα τελεί υπό αναστολή δυνάμει του άρθρου 96 της Συμφωνίας Κοτονού ε, είναι κάτι που γελιοποιεί το Κοινοβούλιο. Δεν δείχνουμε ότι είμαστε υπεύθυνοι και ότι ακολουθούμε τις αρχές μας. Αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ψηφίσαμε ακόμα στην Επιτροπή Ανάπτυξης πάνω σε αυτό, αλλά νομίζω ότι μπορούμε τελικά να πετύχουμε υποστήριξη στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε Σκαντέκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ τον Βιτσέντζο για το έργο του. Νομίζω ότι ήδη είχαμε παρόμοια προβλήματα σε άλλε συμφωνίε, όπω η Μαυριτανία. Σα μην τα βάζουμε όλα στα δύο τσουβάλι. Είναι σημαντική αυτή η έκθεση και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Μαδαγασκάρη. Για μα ειδικά τα παραγαδιάρικα της Ρελνιό, που είναι υπερπόντιο διαμέρισμα της Γαλλίας, ε, πραγματοποιεί 70% των ε, λευμάτων στα χωρικά ύδατα της Μαδαγασκάρης. Και με τους δορυφορικούς ελέγχους και τις δηλώσεις ε, εισόδου-εξόδου εξασφαλίζονται ελέγχη και βιώσιμη εκμετάλλευση των αλλιευμάτων, των χωρικών υδάτων της από τους αλλοδαπούς αλλιευτικούς στόλους. Επίσης, αυξήθηκε και η τομεακή ενίσχυση ώστε να συνεχιστούν ε, οι υγειονομικές, ε, οι υγειονομικοί έλεγχοι και γενικώ η δορυφορική επιτήρηση. Έχουμε αύξηση των αλλιευμάτων με αύξηση της χωρητικότητας. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι αυξήθηκε και η χρηματοοικονομική αντιπαροχή από τους ε, εφοπλιστές. Ε, λογικό είναι άλλωστε, αυξάνονται τα αλλιεύματα, αυξάνεται και η χρηματική αντιπαροχή. Βέβαια, ε, εξασφαλίζεται μία συνέχεια και συνέπεια της διαχείρισης μεταξύ της συμφωνίας και Τη περιφερειακή οργάνωση που είναι αρμόδια για θέματα τη ελία. Εγώ θα ήμουν υπέρ της ε, στήριξης αυτής τη συμφωνία, γιατί όπω είπε και η Ζαμπέλα, τον ε, Απρίλιο θα ε, διεξαχθούν εκλογέ. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη συνέχεια τη Ελληνική Συμφωνίας. Η Μαδαγασκάρη σημείωσε σημαντική πρόοδο, ακολουθώντα κατά γράμμα το φιλοπορία για τη διέξοδο από την κρίση. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή γίνονται πολλές προσπάθειες πρόοδου στη Μαδαγασκάρη. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή και με την έγκριση της συμφωνίας ε, δίνουμε και κάποιες οικονομικές διεξόδους στη Μαδαγασκάρη χάρη στην ατομιακή ε, ενίσχυση που προβλέπει η Ελευτική Συμφωνία. Επαναλαμβάνω, η συμφωνία είναι σημαντική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Μαδαγασκάρη. Και το γεγονός ότι επίκυνται ε, σύντομα εκλογές είναι πολύ καλό μαντάτο. Πιστεύω ότι ήδη από τώρα θα πρέπει να κυρώσουμε αυτή την αλληλευτική συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Καντέκ. Κυρία Φράγκα. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ριμπελίνη για την έκθεσή του. Να πω ότι αν αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα που έχει η κυρία Λέβεν με το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα να πω το εξή. Η πολιτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Μαδαγασκάρη και ο δικός χάρτης δίνουν πολύ θετικά μηνύματα σε ένα οδικό χάρτη μιας χώρας που έδειξε επιθυμία και βούληση να σταματήσει το αυταρχικό καθεστώ και να οργανώσει δημοκρατικές εκλογές. Δόθηκαν πολλά θετικά μήνυματα και καλό θα ήταν να τα συνεχίσουμε με την έγκριση μεταξύ άλλων της συγκεκριμένη αλληλευτικής συμφωνίας. Και από ό,τι ξέρω, χωρί κανένα πρόβλημα πέρασε το θέμα από τις υπηρεσίε Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η Γενική Διεύθυνση ε, Αλίας ε, είπε ότι είναι σημαντικό αυτό το μήνυμα που θα δώσει η Αλληλευτική Συμφωνία προς τη Μαδαγασκάρη και θα δείξει εμπράκτος την υποστήριξη που προσφέρουμε στην ε, χώρα αυτή για να εξέλθει από την πολιτική κρίση. Και στο Συμβούλιο, με εξαίρεση τη Σουηδία, ενέκρινε την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας. Θα πρέπει να το πούμε και αυτό θεωρώ ότι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνταχθεί με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα, υποστηρίζοντας αυτή την ληφτική συμφωνία και δίνοντας ένα θετικό μήνυμα. Εκτός βέβαια και γίνει καμία καταστροφή και μια πολιτική τροπή απρόβλεπτη, κάτι που απευχόμαστε. Τότε μπορεί να, να στείλουμε ακόμα και τις ενισχύσεις. Πάντως άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή την ε, στην ε, γνωμοδότηση κυρία κυρίας Σελόβιν, παρόλο που δεν έχει εγκριθεί ακόμη στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Ε, αναγνωρίζει κύριε ότι ακόμη και στο θέμα των καρχαριών έγινε κάποιο πρόοδος. Και πιστεύω ότι και το πρωτόκολλο καλό θα ήταν να επιδοκιμαστεί. Μετά το λιμάνι της ε, Βικτόρης Σεϊχέλες, η Μαδαγασκά, είναι το, πιο σημαντικό, το δεύτερο πιο σημαντικό λιμάνι για τα θυναλιευτικά. Και μετά τις Αιχέλες, το δεύτερο μεγαλύτερο λιμάνι για τα θυναλιευτικά είναι το λιμάνι της Μαδαγασκάρης. Και μάλιστα αξιοποιείται ιδιαίτερα και από τη μεταπητική μηχανία. Όλα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία και για τον αλληλευτικό κλάδο και το δικό μας και της Μαδαγασκάρης. Πιστεύω ότι η Επιτροπή Αλίας καλό θα ήταν να υποστηρίξει, να υπερψηφίσει την έκθεση. Συμφωνώ απόλυτα με τη θέση του Συγγετού του κ. Ριβελίνη. Ευχαριστώ κυρία Φράγκα. Κυρία Γκαρθία. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να πω εν συντομία ότι όλες οι συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αλληλευτικές συμφωνίες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν θα έπρεπε να έχουν ε, με εξαίρεση τις ελευθερικές ποσότητες θα έπρεπε να έχουν το ίδιο ενδιαφέρον και να δείχνουν τις ίδιες ε, αντιμετώπισης. Είναι σημαντική αυτή η συμφωνία, αλλά εξού σημαντική είναι η συμφωνία και με το Μαρόκο. Ενώ τη συμφωνία με το Μαρόκο την ε, απορρίψαμε. Και στην τελευταία συνεδρίαση που είχαμε και ελπίζαμε ότι θα ήταν καρποφόρα, η αποτυχία ήταν παταγώδης και οι ε, εφαπλιστές και οι αλλοίς που κανονικά αλλοίευαν στα χωρικά του Μαρόκου έχουν μείνει με δεμένα χέρια. Θέλουμε μια συνέπεια στην εξωτερική μας αλληλευτική πολιτική όλοι είμαστε υπέρ της μεταχείρισης και όλοι είμαστε υπέρ της, ε, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αναγνώρισης των συστάσεων ε, της ε, Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας, αλλά φαίνεται ότι εδώ δεχόμαστε την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση αυτά που λέει η έκθεση που διάβασα σύντομα. Εγώ συμφωνώ να υπογραφεί το πρωτόκολλο, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ασκήσει πιέσει. Το εξάμεινο είναι αρκετό διάστημα για να καταλάβει η κυβέρνηση ότι αυτή η ρήτρα, ακόμη και δεν τη τηρήσει, γιατί εγώ α, κατάγομαι μια χώρα που οι ρήτρε αυτές δεν τηρούνται για πάρα πολύ καιρό. Παρ' όλα αυτά λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αποποιηθεί τις θεμελιώδεις της αξίες και αρχές. Και δεν πρέπει ε, στις αλληλευτικές συμφωνίες να παραγωνίζουμε πλήρως ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα τα πρωτόκολλα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τη ρήτρα σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού των εργαζομένων των, ε, ε, των δικαιωμάτων των εργαζομένων με βάση τις προδιαγραφές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εργασίας και σεβασμός της δημοκρατίας. Δεν ε, θα πρέπει να υπογράφουμε τις αλληλευτικές μας συμφωνίες ερήμην όλων αυτών των θεμάτων και των αρχών που αποτελούν θεμελιώδεις αξίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα θεωρούμε ότι είμαστε καταπληκτικοί και πολύ συνεπείς. Με ανησυχούν όλα αυτά. Και για τον ίδιο λόγο και με το ίδιο σκεπτικό και μάλιστα για ίσονο σημασία θέματα και θέματα εδαφικότητας ε, δεν υπογράψαμε τη συμφωνία, την αντίστοιχη συμφωνία με το Μαρόκο, παρόλο που και εκεί υπήρχε επίγουσα κατάσταση και έπρεπε να την είχαμε υπογράψει. Ευχαριστώ κυρία Γαρσία. Κύριος Βεσέρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε. Αυτή η συμφωνία με τη Μαδαγασκάρη είναι έξοχη συμφωνία επί της ουσίας όσον αφορά τις διατάξεις που περιέχει είναι μια συμφωνία υποδειγματική θα έλεγα με την επιφύλαξη βέβαια της ρήτρα ε, εμπιστευτικότητας που ανέφερε η συνάδελφος, η Ιζαμπέλα. Αυτό είναι το ένα. Αλλά δεν μπορούμε να αποσυνδέσουμε, να διαχωρίσουμε μια έξοχη συμφωνία ε, με τις τεχνικές διατάξεις από το πλαίσιο το πολιτικό. Κατανοώ τα επιχειρήματα του Αλέ και του εισηγητή. Δηλαδή, δίνοντας αμέσως τη συμφωνία μας, ενθαρρύνουμε μια μεταβατική περίοδο προς τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Αλλά τι μας υποχρεώνει να προχωρήσουμε τόσο γρήγορα, τι μας υποχρεώνει. Είναι συγκεχημένη η κατάσταση, δεν έχουμε εγγυήσει από αυτή την πλευρά και τα πολιτικά μηνύματα που θέλουμε να στείλουμε κινδυνεύουμε να είναι θολά, συγκεχημένα. Μήπως αντιθέτως το καλό πολιτικό μήνυμα θα ήταν να είμαστε συνετοί, να δείξουμε στεναρότητα, σταθερότητα, λέγοντας ότι αναμένουμε, περιμένουμε, είμαστε έτοιμοι να επικυρώσουμε αυτή τη συμφωνία σε όλες τις διαστάσεις υπό τον όρο ότι απαραίτητο θα πρέπει να διαργηθούν σωστά οι εκλογές, να γίνουν σεβαστές οι δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα να δριωθούν και το κράτος δικαίου να είναι προτεραιότητα για τη Μαδαγασκάρη. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε από αυτή την έποψη. Αντιθέτως, αυτή η σταθερότητα στην στάση μας δείχνει ότι δεν εξετάζει χωριστά τις αρχές με τα τεχνικά ζητήματα, όλα είναι ένα σύνολο. Έχουμε κάθε συμφέρον να καθυστερήσουμε την ψηφοφορία, δεν χρειάζεται να περιμένουμε πολύ χρόνο, τον Απρίλιο, τον Μάιο θα γίνει ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών στη Μαδαγασκάρη. Ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εκτυλιχθούν τα πράγματα. Ας είμαστε συνετοί. Αρχή της πρόληψης από τη δημοκρατική πλευρά και όχι μόνο από πλευράς αλληλευτικής ε, δυνατότητας, αλληλευτικού δυναμικού. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε τους ευρωβουλευτές που θέλαν το λόγο. Δεν ξέρω αν ο κύριος Σεσάριο θέλει το λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους. Καταρχάς θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την έκθεσή του που είναι πολύ θετική, που επικεντρώνεται επί των βασικών στοιχείων και εμείς μετά από την παρούσα συζήτηση θέλουμε να διακρίνουμε τα δύο μέρη, να τα διαχωρίσουμε, υπενθυμίζοντας ότι η διαπραγματευτική μας διαδικασία εξετυχθεί σε στενό συντονισμό με την εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως καθ' όλη τη διάρκεια των διαδικασιών. Και είχαμε και επαφές με την αντιπροσωπεία της Μαδαγασκάρης. Ποτέ ε, δεν λησμονήσαμε την πολιτική κατάσταση που επικρατεί στη Μαδαγασκάρη. Το ίδιο έκανε και το Συμβούλιο όταν έδωσε την εντολή. Όσον αφορά την αλληλεία, υπογραμμίστηκε κάτι που επαναλαμβάνω. Εμπεριέχονται στοιχεία θετικότατα, σύμφωνα με την μεταρρύθμιση, αύξηση της τομεικής υποστήριξης, ηλεκτρονική ανταλλαγή στοιχείων, υπάρχουν διάφορες πτυχές η βελτίωση της διαχείρισης των πόρων και αναφέρομαι στον περιορισμό ε, της ε, αλίας των ε, σκυλόψαρων, των καρχαριών, που είναι κάτι καινοτόμο όσον αφορά την περιφερειακή διαχείριση, ε, όσον αφορά την αλληλεία στον Ειδικό ωκεανό, πολλά θετικά στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όσον αφορά τις πολιτικές πτυχές, σεβόμαστε απόλυτα τι απόψει που εξεφράστησαν από τα αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου, αυτό μπορούμε να διαπιστώσουμε ακόμα μια φορά όμως, ε, ε, ε, ενώ είμαστε επαφή με την εξωτερική υπηρεσία του συναδέλφου, υπάρχουν πρόσφατε θετικέ εξελίξει, θετικότατε. Τα, τα μάθαμε αυτά τι πρόσφατε ημέρε. Η Βαρόνια Άστον μα ενημέρωσε στι 19 Ιανουαρίου σχετικά με αυτό. Υπάρχουν σημάδια από πλευρά του Προέδρου του και του πρώην Προέδρου ότι δεν θέλει να είναι ξανά υποψήφιο στι προεδρικέ εκλογέ. Άρα βλέπουμε θετικές εξελίξεις όσον αφορά την εφαρμογή του χάρτη πορείας. Είμαστε ε, αισιόδοξοι. Θα ήταν θετικό μήνυμα πλευρά Ευρωπαϊκή Ενώσεω η κύρωση τη συμφωνία και γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η τομική στήριξη για την Μαδαγασκάρη όσον αφορά του διαθεσίμου πόρου. Λοιπόν, θα θέλαμε να επικυρωθεί το ταχύτερο δυνατόν αυτή η συμφωνία. Δεν θα μακρηγορήσω επί των άλλων περιφερειακών και ελευτικών πτυχών. Είναι μια συμφωνία που αποτελεί ένα τμήμα του δικτύου συμφωνιών των περιφερειακών του Ινδικού ωκεανού και εντάσσεται όπως ήδη αναφέρθηκε, τέλεια στο πλαίσιο της, ε, του πλαισίου διαχείρισης Επιτροπής του Ινδικού Οκεανού. Όσον αφορά τη ρήτρα εμπιστευτικότητα, ε, ήδη χτες προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε το θέμα στην Επιτροπή Ανάπτυξης. Η ρήτρα αυτή αντικατοπτρίζει άλλα νομοθετικά μέσα όπως παραδείγματος τον κανονισμό για το VMS ή διεθνείς κανόνες όπως το θέμα της εμπιστευτικότητας, ε, εμπιστευτικότητας της Επιτροπής του Δικού Ωκεανού. Υπάρχει κάποια αμφισημία, αμφιβολία όσον αφορά τη διατύπωση του κειμένου. Τι θέλαμε, θέλαμε να προστατεύσουμε τις εμπορικές πτυχές. Αυτό ε, θέλαμε να καλύψουμε. Αν υπάρξει ανάγκη να, το, να επεξηγήσουμε αυτή την προσέγγιση. Σίγουρα είμαστε στη διάθεσή σα ε, να ετοιμάσουμε μια μεικτή επιτροπή και να δούμε ποιο κείμενο, ποιο κείμενο θα μπορούσε να είναι πιο ενδεδειγμένο και θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε μελλοντικέ συμφωνίε. Διότι η ουσία ποια είναι. Θέλουμε στον ειδικό ωκεανό κυρίω θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την πειρατεία, θέλουμε να στηρίξουμε την ασφάλεια. Και τα ευαίσθητα εμπορικά στοιχεία εξασφαλίζοντα την πρόσβαση στα στοιχεία και από πλευρά των κυβερνήσεων και δικήσεων και από πλευρά των επιστημόνων που χρειάζονται αυτά τα στοιχεία. Θα σταματήσω εδώ κύριε Πρόεδρε. Α ελπίσουμε ότι θα μπορέσει να εγκριθεί η συμφωνία από το Κοινοβούλιο διότι αν α, απορριφθεί δεν θα είναι πολύ θετικό το μην θα στείλουμε στην Μαδαγασκάρη και θα αμφισβητηθούν στις διαπραγματεύσεις όλα τα θετικά συμφωνία, τα αλληλευτικά, τα οποία έχουμε συμπεριλάβει ε, όσον αφορά ε, τη, μείωση της αλίας των καρχαριών ε, που νομίζω ότι είναι μια εξέλιξη πάρα πολύ θετική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Τσέζερη. Ο κύριος Ριβελίνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για όσα είπαν για μένα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με τον κ. Λαβίν και με την ε, Επιτροπή που έδειξε ανοιχτή ε, για να υποβληθεί μια τροπολογία που θα, κατά κάποιο τρόπο θα αναδιατυπώνει και θα βελτιώνει, ε, θα καθησυχάζει τις ανησυχίες. Να μελετήσουμε τις τροπολογίες που μπορούν να διευκρινίσουν, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το άρθρο 11. Όσον αφορά τις πολιτικές πτυχές, και αυτά που είπε μόλις τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας κάνουν να καταλάβουμε ότι έγιναν διπλωματικές διαπραγματεύσεις ε, και οδήγησαν σε αποτελέσματα διπλωματικές επαφές. Εμείς όλοι οι βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου εκπροσωπούμε τα δικαιώματα που από τη δημοκρατία. Ε, όλα αυτά που ανέφερε και Λουβίν, κανείς ε, δεν θέλει να υπάρξει επαναχώρηση, αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε με προσοχή ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι η διπλωματική στάση ε, που δίνει καρπούς ε, και θα ζητούσα από τους συναδέλφους να ψηφίσουν, να εγκρίνουν την έκθεση. Ε, βέβαια χρειάζεται για το άρθρο 11 μια τροπολογία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω ο κύριος Τσέσσερι να προσθέσει κάτι. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που παίρνω ξανά το λόγο. Θα ήθελα να διευκρινίσω όμως κάτι, διότι ίσω δεν έγινα, δεν υπήρξα σαφέστατο. Ποια είναι η θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πιστευτικότητα. Είμαστε στη διάθεσή σα να εργαστούμε επί του παρόντο κειμένου, επί αυτή τη βάση. Δεν προτείνουμε μια τροπολογία όσον αφορά το παρόν κείμενο. Είμα, μπορούμε σε τεχνικό επίπεδο να επεξεργαστούμε, να εξηγήσουμε αυτό το σημείο που έχει αυτή τη διατύπωση σε επίπεδο μεικτή επιτροπή με του φίλου μα από τη Μαδαγασκάρη όταν θα συνεδριάσουμε και στο μέλλον για διαφορετικές συμφωνίες σίγουρα θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε σαφέστερα την έννοια που προσπάθησα να εξηγήσω σήμερα εδώ. Δηλαδή η προστασία των εμπιστευτικών στοιχείων που είναι εμπορικά ευαίσθητα. Θέλω να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν προτείνει ε, να τροποποιηθεί το κείμενο, να διαπραγματευτούν το κείμενο. Προτείνει να το διευκρινίσουμε σε τεχνικό επίπεδο στην Μικτή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε η κυρία Λάβιν πρότεινε να μην ε, δώσουμε συνέχεια στο θέμα, αλλά υπήρξαν πολλές παρεμβάσεις ε, που ακολούθησαν ε, την αντίθετη γνώμη. Η πλειοψηφία τάστη υπέρ της συνέχισης και στις 29 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, θα λήξει η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Αν έχουμε ξαφνικές εξελίξεις, ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε και τον τρόπο δράση. Πάντω, συνεχίζουμε και προθεσμία 29 Ιανουαρίου στι 12 το μεσημέρι. Προχωράμε στο σημείο 12 τη ημερήσια διάταξη. Την τροποποίηση του κανονισμού 1100 του 2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού. Στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου έγινε μια παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σήμερα θα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την εισηγητριά μας, την κυρία Λόβιν. Έχετε το λόγο κυρία Λόβιν. Thank you very much. Ευχαριστώ πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή είναι πολύ σημαντική στιγμή εδώ για μένα στην Επιτροπή Αλίας γιατί το ενδιαφέρον μου για την ε, αλληλεία ε, δημιουργήθηκε όταν ε, κατάλαβα πως έχει κατάσταση για το ευρωπαϊκό χέλι. Ε, ήδη από το 2003, δηλαδή πριν από μια δεκαετία. Πριν από δέκα χρόνια ήμουν δημοσιογράφος σε ένα σουηδικό περιοδικό και έλαβα ένα ανακοινωθέν τύπου από το Σουηδικό Συμβούλιο Αλίας που έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήθελε να κλείσει την ε, δυνατότητα αλίευσης για τη Σουηδία για το χέλι, γιατί το ευρωπαϊκό χέλι βρισκόταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ήταν σε κατάσταση κατάρρευση στο απόθεμα. Πριν από 10 χρόνια, βεβαίω, η κυβέρνησή μου διαμαρτυρήθηκε και το ίδιο έκαναν και οι υπόλοιπε κυβερνήσει. Γιατί το ευρωπαϊκό χέλι είναι κοινό απόθεμα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πιστεύουν ότι στη χώρα τους το ε, χέλι τους είναι ε, Ιρλανδικό, Ιταλικό, Γαλλικό, Εθνικό τέλος πάντων. Δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό χέλι και ένα, ένα απόθεμα ευρωπαϊκού χελιού που είναι κάτι πολύ συμβολικό ε, για την Επιτροπή μας. Όλα τα ευρωπαϊκά χέλια ε, αναπαράγονται στα μέσα του, στην, κάπου στον Ατλαντικό και μετά πεθαίνουν. Κάποια μικρά έρχονται με το ρεύμα προς τις ευρωπαϊκές ακτές, κάποια πάνε προς τα νότια της Ευρώπης, κάποια προς τα βόρεια κάποια μικρά ηχθίδια περνούν από τη Γιβραλτάρ, α πούμε, στη Μεσόγειο και πάνε στην Ιταλία. Ή και αλλού παντού στην Ευρώπη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά πάντα μιλούμε για το ίδιο απόθεμα. Ήδη λοιπόν από το 2003 είχε μειωθεί κατά 99% η, ε, ο γόνος του χελιού. Τα χέλια μεταναστεύουν σε γλυκά νερά, σε λίμνες, έχουν δηλαδή αντεστραμμένο κύκλο ζωής από το Σολομό, γεννιούνται δηλαδή σε αλμυρό νερό, αλλά ζουν σε γλυκό νερό. Στη Βόρεια Ευρώπη μπορεί να ζήσουν μέχρι και 30 χρόνια πριν μεταναστεύσουν ε, μεταναστεύουν συνήθως όταν έχει πανσέλινο και εκεί ε, ε, μεταναστεύουν, αναπαράγονται και πεθαίνουν πάλι πίσω στον Ατλαντικό. Μπορεί να μην υπάρχει βεβαίως τόσο τεράστια μείωση των ασημόχελων και των κυτρινόχελων όπως υπήρχε πριν από 10 χρόνια, αλλά τα κίτρινόχελα βρίσκονται κυρίως σε γλυκά νερά, εκεί ζουν. Ε, υπάρχουν λοιπόν πολλές φάσεις στον κύκλο ζωής για, τον, ε, ε, για τα χέλια. για τα σημόχελα, τα κιτρινόχελα, τα αμόχελα, όλα αυτά είναι το ίδιο απόθεμα, είναι το ευρωπαϊκό χέλι. Όταν λοιπόν ανέλαβα εγώ ως εισηγήτρια για την λισαβονοποίηση του κανονισμού για τα χέλια. Πραγματικά ήταν κάτι πολύ ενδιαφέρον και το ανέλαβα με χαρά. Γιατί για μένα αποτελεί μυστήριο από το 2003 πώς θα επιτρέψουμε πώς θα, τι θα κάνουμε, πώς θα διαχειριστούμε την, α, ε, ε, την αλλιεύση αυτού του, πολύ, που, αυτού του αποθέματος που βρίσκεται σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Ε, είχαμε πει ότι δεν μπορούμε να περιορίσουμε την αλληλεία μας. Έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις ήδη και από παλιά. Το 2007 τελικά όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης συμφώνησαν σε ένα σχέδιο ανάκτησης του χελιού και αυτό ακριβώς έχουμε τώρα εδώ, για, στα πλαίσια πάντα της λισαβονοποίησης. έχει κάποιες ε, διατάξεις που λένε ότι τα κράτη-μέλη θα υποβάλουν μια αξιολόγηση για το πώς προχωρεί το πράγμα από το 2007 και αυτό πρέπει να το έχουν ήδη κάνει πέρσι. Η Κομισιόν θεωρητικά θα υποβάλει μια νέα πρόταση με βάση αυτές τις αξιολογήσεις. Ποιος είναι τώρα ο στόχος αυτού του σχεδίου ανασύστασης. Ε, ο στόχος είναι αρκετά παράξενος. Λέει ότι όλα τα κρατη θα πρέπει να προσπαθήσουν ε, ώστε το 40% ενός ε, υγιούς αποθέματος χελιού θα πρέπει να επιτρέπεται να μεταναστεύει και να, ε, να αναπαράγεται of the biomass of silver eel. στη θάλασσα των Σαργασών. Με βάση βεβαίως και τις ε, συνθήκες τις οποίες ε, ισχύουν για αυτό ακριβώς το ικανό κομμάτι του αποθέματος. ελπίζω να έχετε καταλάβει τι εννοώ. Έχω δει έχω διάφορες αξιολογίες των κρατών μελών και είναι σαφές ότι τα κράτη-μέλη έχουν τελικά διαφορετικές, διαφορετικό ορισμό αυτού του τι σημαίνει το 40% του, της βιομάζας του ασημόχελου πάντα μέσα σε κάποιες ε, κανονικές συνθήκες. Είναι δύσκολο λοιπόν να υπολογιστεί αυτό και υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να υπολογιστεί, αλλά κανένας από όσους είδα τουλάχιστον εγώ δεν με καθησύχασε για το ότι τα πράγματα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια, αν δείτε πώς ε, επετεύθη ο στόχος αυτός από τα κράτη-μέλη, μάλιστα η ISIS ποτέ δεν έχει αξιολογήσει το στόχο αυτό. Η ISIS λοιπόν λέει σαφώς ότι το 40% της μετανάστευσης, της διαφυγής δεν ήταν δική τους ε, σύσταση. 50% μπορεί να ήταν λίγο πιο ε, συναφές με τις δικές τους συστάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτός είναι πολιτικός στόχος. Έχω δει το τι έχουν επιτύχει τα κρατημέλη μέχρι τώρα. Υπάρχουν διάφορες μελέτες, εκθέσεις, ε, καθόλου εναρμονισμένες μεταξύ τους. Οι εκθέσεις έχουν γίνει με τελείως διαφορετικό τρόπο αναχώρα. Αυτό που σας λέω ίσως να μην είναι απόλυτα σωστό, γιατί υπάρχουν και κάποιες άλλες ε, γλώσσες. Καταλαβαίνω εγώ γαλλικά, γερμανικά, λίγα ιταλικά, λίγα ισπανικά, λίγα πορτογαλικά, αλλά... Ε, εντάξει, ίσω να μην έχω ερμηνεύσει απόλυτα σωστά και δεν έχω διαβάσει βεβαίω και τα πάντα από την αρχή μέχρι το τέλο αλλά ε, με τα δανέζικα και τα σουηδικά και τα αγγλικά τα πάω καλά και τα περισσότερα από όσα διάβασα ήταν στα αγγλικά. Οπότε από ό,τι έχω καταλάβει από τα κράτη-μέλη, δεν υπάρχει κανένα από τα κράτη-μέλη που να έχει πετύχει το συνολικό στόχο του 40% διαφυγής του ασημόχελου σε σχέση με την ε, καλύτερη δυνατή αξιολόγηση, εκτίμηση της ε, θεωρητικής διαφυγής του αποθέματος ασημόχυλου. Στη Σουηδία είχαμε 25% ποσοστό διαφυγής συμπεριλαμβανομένης και της ε, ε, ανασύστασης του αποθέματος και αυτό είναι σημαντικό. Το Βέλγιο έχει φτάσει το 20%, η Τσεχία, η Σλοβακία 16 με 22, η Δανία αν έχω διαβάσει καλά είναι περίπου στο 11% αν δεν κάνω λάθος, η Πολωνία 4%, Ενωμένο Βασίλειο περίπου 25%, Ισπανία περίπου στο 15% και τα λοιπά. Η Γερμανία 25 με 30, η Ιταλία 16%. Πορτογαλία, η Πορτογαλία λέει ότι δεν μπορεί να το υπολογίσει και τα λοιπά η Ιρλανδία είναι πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα, γιατί είναι η μόνη χώρα, το μόνο κράτος μέλος, που έκλεισε την ελεία του. Εντελώς. Και ούτε καν η Ιρλανδία δεν πέτυχε τον στόχο του 40%. Βρίσκεται περίπου στο 24 ε, με πάνω από 40 σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι λίγο περίεργο να διαβάσει κανείς και να κατανοήσει όλες αυτές τις αξιολογήσεις γιατί δεν έχουν γίνει όπως σας είπα με έναν εναρμονισμένο ομοιογενή τρόπο. Είναι σαφές όμως ότι η ΆΙΣΕΣ ποτέ δεν είπε ότι το 40% διαφυγής είναι καλός στόχος ή ότι είναι αρκετό και τα κράτη-μέλη από ό,τι έχω διαβάσει εγώ δεν τον έχουν επιτύχει. Μπορεί κανείς να πει βέβαια ότι ε, εντάξει, αλλά από το 2007 ξεκίνησε να τρέχει αυτό. Ναι, αλλά εγώ σας είπα ότι αυτό το, αυτή τη συζήτηση την κάνουμε εδώ και 10 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Το 2003 η Κομισιό ήθελε να κάνει κάτι. Ήδη από τότε. 10 χρόνια μετά είμαστε πάλι εδώ και τα κράτη-μέλη έχουν αποδειχθεί α, ε, αργά στην όλη ε, εφαρμογή της διαδικασίας. Δεν ξέρω αν έχετε αντίτυπο των ε, συστάσεων της ISIS. Ένας από τους λόγους που ήθελα να καθυστερήσω την περαιτέρω συζήτηση για την έκθεση μαζί σας είναι γιατί ήξερα ότι θα υπάρξει νέα σύσταση από την ISIS ε, το Νοέμβριο. Μετά δηλαδή από την τελευταία μας συζήτηση. Αυτή η σύσταση πρέπει να την έχετε λάβει. Λέει αυτά που πρέπει. Το απόθεμα χελιού εξεκολουθεί να, να μειώνεται το 2011. Έχει, έχουν μειωθεί η, η τάση διαφυγής από το, στο 5%. Για τα, για τα γυαλόχελα δεν βλέπουμε δυνατότητα ανασύστασης. Το γελόχυλο, το αμόχυλο και το ασημόχυλο βρίσκονται σε ιστορικό χαμηλό. Το απόθεμα βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το 2007 το, ε, το χέλι μπήκε στο παράρτημα 2 της ΣΑΙΤΕΣ που δεν θεωρείται βέβαια ε, είδος προς εξαφάνιση, αλλά ε, καλό θα ήταν να μην γίνεται αλίευσή του έτσι ώστε να επιβιώσει το είδος η κατηγοριοποίηση ε, ξεκίνησε να ισχύει το 2009, το ε, χέλι μπήκε τον ε, Σεπτέμβριο του 2008 ως, κρίσιμο, ως απόθεμα σε κρίσιμη κατάσταση, στον κόκκινο δηλαδή κατάλογο. Και ήθελα να πω ότι ο κατάλογος σε site στο παράρτημα 2 υπάρχει γιατί η μόνη πρόταση για καταχωρήσεις ήταν για το παράρτημα 2, αλλά επιστημονικά θα μπορούσαν οι καταχωρήσεις να γίνονται και στο παράρτημα 1. Το παράρτημα 1 απαγορεύει οποιαδήποτε εμπορική διαδικασία είτε με ζώντα είτε με νεκρά δείγματα αυτού του είδους. Ξέρω ότι υπάρχει συζήτηση που γίνεται ώστε το χέλι να μπει στο παράρτημα 1. Φανταστείτε λοιπόν τι θα σήμαινε αυτό για την αλίευση χελιού. Πάμε τώρα στην ανασύσταση του αποθέματος που σημαίνει ότι ε, ε, αλλιεύουμε σε μία λεκάνη μικρά ηχθίδια για και τα μεταφέρουμε σε ένα άλλο σημείο όπου υπάρχουν λιγότερα χέλια και υπάρχει ένα οικότοπος όπου θεωρούμε ότι θα μπορούσε το χέλι να αναπτυχθεί. Αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με τον κανονισμό για την ανασύσταση του αποθέματος χελιού. Παρόλα αυτά, το 2010 η ΆΙΣΕΣ για πρώτη φορά ανέφερε ότι το γελόχελο και το, απόθεμα επανασύσταση, το πρόγραμμα επανασύστασή τους μάλλον δεν θα ενισχύσει την, ουσιαστικά το πρόγραμμα ε, ανασύστασης του ευρωπαϊκού χελιού. Και δεν υπάρχει και απόδειξη για το ότι όντως ε, η ανασύσταση του γελόχελου βοηθάει την ανασύσταση του ευρωπαϊκού χελιού. Αυτό ήταν, ε, ήταν σημαντικό όταν, ε, όταν ε, εκδόθηκε και βεβαίως οδήγησε και την Κομισιόν στο να αναθεωρήσει όλα τα σχέδια ανάκτησης των κρατών μελών, γιατί πολλά εξ αυτών και το πολωνικό και το σουηδικό ακόμα και το τσεχικό, πολλά λοιπόν από αυτά βασίζονται στο πρόγραμμα ανασύστασης για την επίτευξη αυτού του στόχου του 40%. Εγώ έθεσα ένα ερώτημα στην Κομισιόν το 2011 και ζητούσα αν μπορεί να γίνει κάτι ώστε να επιταχυνθεί όλη η διαδικασία και να δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρξει κάποια εγγύηση για την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Αποθέματος Χελιού, όπως ζητάει και η ISS. Ε, μου απάντησε λοιπόν, ε, έλαβα μάλλον μια απάντηση από την κυρία Δεμανάκη που έλεγε ότι τα κρατημέλη έχουν υποβάλει τα σχέδια διαχείρισης τους χωρίς ε, ε, καθυστέρηση. Ε, κάποια βέβαια βρισκόνταν και σε μια αλφα καθυστέρηση κάποιων μηνών ή ενό ή δύο ετών. Ε, οπότε τώρα η ενος η δυο ετων ε πρέπει να αξιολογήσει αυτά τα προγράμματα. Βεβαίως η Κομισιόν δεν ε, αποκλείει τα μέτρα τα επίγουσας κατάστασης σε σχέση με την αλλιεύση του χελιού. Και αυτό έγινε τον Μάιο του 2011, δηλαδή σχεδόν πριν από δύο χρόνια. Οπότε τα πράγματα πραγματικά κινούνται πάρα πολύ αργά. Και το μόνο που είναι σίγουρα σαφές είναι ότι η ISIS δίνει τις συστάσεις της κάθε χρόνο και λέει ότι θα πρέπει η ανθρωπογενής θνησιμότητα των χελιών να μειωθεί όσο δυνατόν περισσότερο ώσπου να φτάσει σε μηδενικό επίπεδο έτσι ώστε να μπορέσει να αυξηθεί το απόθεμα. Αυτό δεν συμβαίνει προς το παρόν. Τώρα θα κάνουμε μια συζήτηση εδώ στην Επιτροπή και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις σας για το τι θα πρέπει να κάνουμε. Έχουμε και την έκθεση ευθυγράμμισης. Η Κομισιόν προτείνει κάποιες μικρές αλλαγές για τις κατεξιότητες πράξεις. Να το δεχτούμε και να κάνουμε απλώς μια ευθυγράμμιση. Να κάνουμε τροποποίηση της έκθεσης της ίδιας. Του κανονισμού μάλλον ε, που Νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί περιλαμβάνει τόσα στοιχεία που δεν έχουν αξιολογηθεί σε επιστημονικό επίπεδο, ούτε τα μέτρα ανασύσταση έχουν αξιολογηθεί, ούτε ο ίδιος ο στόχος έχει αξιολογηθεί. Ή θα πρέπει να τραβήξουμε το, να χτυπήσουμε το σήμα κινδύνου τώρα. Υπάρχει μια δυνατότητα η Κομισιόν να εφαρμόσει τέτοια μέτρα επίγουσας ανάγκης, έκτακτης ανάγκης. Στο άρθρο 7 του βασικού κανονισμού λέει ότι, ότι εκεί η Κομισιόν μπορεί να πάρει μέτρα επίγοντα. Αν δηλαδή υπάρχει απόδειξη άμεση σοβαρής απειλής των θαλάσσιων πόρων ή του θαλάσσιου οικοσυστήματος που απορρέουν από αλλιευτικές δραστηριότητε και χρειάζονται άμεση δράση. Η Κομισιόν, μετά από αίτημα των κρατών μελών ή από δική της πρωτοβουλία, μπορεί να αποφασίσει να λάβει έκτακτα μέτρα τα οποία δεν θα κρατήσουν πάνω από 6 μήνε. Η Κομισιόν μπορεί να λάβει νέα απόφαση για επέκταση αυτών των μέτρων για άλλο ένα εξάμεινο και όχι παραπάνω. Η Κομισιόν λοιπόν μπορεί να κλείσει την αλίευση χελιού όσο θα αξιολογεί τις εκθέσεις των κρατών μελών και να υποβάλει μια νέα πρόταση με βάση επιστημονικές, επιστημονικά στοιχεία για το πώς θα προχωρήσουμε. με την αλίευση αυτού του είδους ή με την ανασύσταση, εν πάση του αποθέματος, γιατί αμφιβάλλω πάρα πολύ ότι θα μπορούμε να συνεχίσουμε να ε, αλλιεύουμε αυτό το είδος που βρίσκεται σχεδόν υπό εξαφάνιση και με βάση την ε, ε, μεταρρύθμιση της κοινής ελευτικής πολιτικής. Εάν όμως κάτι δεν το αλλιεύουμε, πρέπει να το συζητήσουμε στην Επιτροπή Αλλιείας. Ε, ναι, αλλά αν πρέπει να σταματήσουμε την αλίευση ακριβώς λόγω υπεραλίευσης, προφανώς θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει ανασύσταση του αποθέματος. Και τα, ε, τα κονδύλια ε, θα πρέπει να δοθούν έτσι ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπάρξει ανασύσταση του ευρωπαϊκού χελιού και δεν είναι βέβαια μόνο η αλληλεία που οδήγησε στην κατάρρευση του αποθέματος, αλλά κανένας επιστήμονας δεν μπορεί να μας πει συγκεκριμένα γιατί μπορεί να είναι λόγω της μόλυνσης, μπορεί να είναι λόγω ασθενειών, ζωνώσεων, μπορεί να είναι λόγω της κλιματική αλλαγή μπορεί να έχουν συμβάλει πολλοί παράγοντες, ε, οπότε δεν ε, πρέπει να καταδεικνύουμε με το δάχτυλο μόνο τους αλληλεί που ψαρεύουν το, τα, τα χέλια, αλλά η κατάσταση βρίσκεται σε αυτή την πολύ δύσκολη φάση και πρέπει κάτι να κάνουμε τώρα. Αυτά λοιπόν είναι τα ερωτήματά μου προς εσάς. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε. Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καντέκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ιζαμπέλα. Έξοχη παρουσίαση. Είναι ε, δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τα πάντα. Πράγματι, ο πληθυσμός των χελιών μειώθηκε κατά πολύ εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχουν πολλά αίτια γι' αυτό. Η Σαμπέλα το είπε. Πρώτα απ' όλα η ρήπανση είναι ένα αίτιο. Η αλλαγή του κλίματος επηρεάζουν όλα αυτά τη συμπεριφορά των χελιών, κυρίως τη μετανάστευσή τους από τη θάλασσα των Σαργασών μέχρι τα ευρωπαϊκά ύδατα και είναι στοιχεία πρέπει να ληφθούν υπόψη υπάρχει και κάτι άλλο πολύ σημαντικό στα στοιχεία. Η υπεραλίευση των ε, μικρών ε, χελιών που αλλιεύονται στην επιστροφή τους από τη θάση των αργασών, τα νεογνά προς τα, υδά, προς τα ε, γλυκά ύδατα. Όταν υπάρχει η παραλίευση των νεογνών, των, μειώνεται σημαντικά το απόθεμα. Η ίδια υπεραλίευση των χελιών πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αν και ίσως είναι στοιχείο περιθωριακό. Και κάτι άλλο που πρέπει να λάβουμε υπόψη και δεν το αναφέραμε, ασχολούμαι εγώ προσωπικά για τη Γαλλία, η συνέχεια, η οικολογική, τα εμπόδια μπορούν να αντιμετωπίσουν τα χέλια που πάνε ανάντι στα ποτάμια για να φτάσουν εκεί που ζουν στα αγγλικά ύδατα. Ε, θέλουμε να μειώσουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν για να φτάσουν στην πηγή. Και αν δεν μπορούμε να τα βγάλουμε, βάζουμε ένα είδος κλίμακας για τα ψάρια, όπως βοηθάμε και τους ολομούς, για να μπορούν να πάνε ενάντια στο ρεύμα ε, του ποταμού. Ε, θα πρέπει κάθε κράτος μέλος να εξετάσει αυτή την πτυχή των πραγμάτων. Είναι αρκετά περίπλοκο θέμα, διότι όπως έλεγε οι επιστήμονες δεν συμφωνούν όλοι όσον αφορά τους λόγους για τη μείωση των χελιών και θέτουν διάφορα ερωτήματα και ομολογώ ότι είναι αρκετά περίπλοκο το θέμα του των λεχθέντων πράγματι η μείωση των χελιών κατά την άποψή μου δείχνει είναι ένα σημάδι της δυσλειτουργίας που οφείλεται ήταν στην αλλαγή του κλίματος, στην υπερλίευση, στη μόλυνση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέξουμε όλο ιδιαίτερο τη μείωση. Να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα. Λαμβάνοντα υπόψη αυτά που είπε, βέβαια, θέλουμε να σταματήσουμε τη μείωση. Ε, είναι σημαντική η μείωση στην Ευρώπη. Σε 15 χρόνια μειώθηκε δραματικά αριθμό των χελιών. Αυτά ήθελα να πω. Αυτέ ήταν κάποιε παρατηρήσει που είχα. Θα πρέπει να επεξεργαστούμε την έκθεση και να κάνουμε τα μέγιστα για αυτό το, το, το είδος ίσως να είναι περιθωριακό σε σχέση με άλλα είδη που αλλιεύονται, αλλά είναι ε, σημαντικό σημάδι, μας δείχνει κάτι και πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτή η μείωση. Ευχαριστώ κύριο Σκούν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την κυρία Λεωβίν, που μας περιέγραψε αυτό το, το μυστικό ε, νομίζω ότι ούτε η επιστήμη δεν μπορεί να λύσει το πρόβλημα. Έχει τεράστια, έχει ε, μάλλον πολύ λίγη εμπειρία για το πώς γίνεται η αναπαραγωγή των ε, χελιών και πώς γίνεται και η ανασύσταση, πώς γίνεται η μετανάστευση, πώς έρχονται με το ρεύμα ή ανάντι ή κατάντι, τι γίνεται με το αρμυρό και το γλυκό νερό. και πώς μπορούν να ζήσουν ε, στα ύδατα αυτά για 25 ή 30 χρόνια. Είναι σημαντικό λοιπόν καταρχάς να μελετήσουμε καλύτερα τα επιστημονικά δεδομένα και είναι καλό που τα έχουμε και στα χέρια μας. Να τα δούμε λοιπόν πιο καλά, να δούμε τι διαφορές υπάρχουν, τι λένε όλα αυτά τα πορίσματα της επιστήμης και τι από όλα αυτά μας βοηθά στη δουλειά μας. Γιατί υπάρχει και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και στην εσωτερική αλεία, όχι μόνο από εμπορική πλευρά, αλλά θα πρέπει να μπορούμε να διατηρήσουμε και, το, και την αλληλεία αλλά και το απόθεμα. Ας πούμε δεν έχουμε καμία ένδειξη τώρα για το πώς, τι κατάσταση είναι το, το απόθεμα. Μιλούμε για την αναπαραγωγή, μιλούμε για τα μικρά, τα ηχθίδια, τα χέλια τα οποία έρχονται προς τα ευρωπαϊκά νερά και πώς ε, περνούν ε, από τον Βυσκαϊκό κόλπο. Ε, πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν πώς εξελίσσεται τελικά ένα απόθεμα. Έχει βελτιωθεί η κατάστασή του, έχει επιδεινωθεί, αυτό είναι σημαντικό. Και πέρα από τα τεχνικά μέτρα, έτσι όπως τα περιγράφει και η Κομισιόν στα σχέδια διαχείρισης, θα πρέπει να υπάρχει και η δυνατότητα να υπάρχει αλίευση. και βεβαίως θα πρέπει να μην ε, τίθεται σε κίνδυνο το, ε, το απόθεμα χελιών, να, μην κινδυνεύει από οποιοδήποτε παράγοντα, ε, είτε από, τα, από πουλιά που μπορεί να, το, να φάνε τα μικρά ηχθίδια, είτε από οποιοδήποτε άλλο παράγοντα. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτά τα σχέδια διαχείρισης, ανακράτος μέλος, και νομίζω ότι θα πρέπει και στο μέλλον να επικεντρωθούμε σε αυτό, γιατί από εκεί μπορούμε να εξάγουμε όντω αρκετά συμπεράσματα για το τι γίνεται με το απόθεμα στα εσωτερικά μας ύδατα, πόση αλίευση υπάρχει αυτού του αποθέματο. και επίσης όταν το, μετά από πολλά χρόνια το χέλι θέλει να επιστρέψει στα ύδατα από, από τα οποία ήρθε, θα πρέπει να δούμε πώς γίνεται αυτό έτσι ώστε να μπορέσει το χέλι να φτάσει στα, στην θάλασσα των Σαργασών. Νομίζω λοιπόν ότι αυτός είναι ένας κύκλος που ξεκινάει και κλείνει. Έχουμε τα σχέδια διαχείριση από το 2007, από το 2009. Έχουν εξελιχθεί, έχουν εκπονηθεί από τα κράτη-μέλη. Κάποιοι δίνουν μπόλικα δεδομένα, κάποιοι δίνουν λιγότερα. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να τα μελετήσουμε γιατί ε, αυτά τα αποτελέσματα, ακριβώ επειδή είναι αποτελέσματα πολλών ετών, μπορούν να μα δώσουν πολλέ ε, γνώσει. Προ το παρόν δεν τι έχουμε. Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο θα τα διαχειριστούμε. Νομίζω ότι να βάλουμε τώρα ε, μορατόριο εδώ και κλείσιμο της αλίας δεν είναι ο σωστός δρόμος για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Νίλσον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω σου ειδικά, αφού υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Σίγουρα υπάρχουν εύλογοι λόγοι ανησυχίας ό,τι αφορά την κατάσταση των χελιών. Πριν από μία δεκαετία μας είπατε ότι είχαμε την πρώτη έκθεση για την κατάσταση του αποθέματος χελιού που ήδη έδειχνε μία πολύ σοβαρή κατάσταση. Και αν δούμε τη διάρκεια ζωής ενός χελιού βλέπουμε ότι είναι αρκετά μεγάλη. Και δεν μπορούμε αμέσως να αντιληφθούμε ε, τον κίνδυνο. Γιατί ε, δεκαετία μπορεί να μας φαίνεται μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δεδομένη στη διάρκεια ζωής του χελιού δεν είναι και τόσο μεγάλο. Τώρα, στη Σουηδία ιδιαίτερα στη Νότια Σουηδία, καταναλώνουμε μεγάλες ποσότητες χελιού. Ε, είναι από τις σπεσιαλιτέ μας συνταγές με χέλι και προσπαθούμε τώρα να περιορίσουμε αυτή την κατανάλωση και να πούμε, στο, να πούμε στον κόσμο και να αντιληφθεί, να συνειδητοποιήσει και ο πολίτη ότι θα πρέπει να μειώσει την κατανάλωση χελιού, γιατί είναι απειλούμενο είδο αυτή τη στιγμή το χέλι. Δεν θέλω να επαναλάβω όλες τις εύστοχες ε, ερωτήσεις που υπέβαλε η Ισαμπέλ Λεωαβίν. Φαντάζομαι θα απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα προσθέσω κι εγώ μερικές δικές μου απορίες. Τι γνώμη έχετε για το υπάρχον σχέδιο διαχείρισης. Θα επιτρέψει αυτό το σχέδιο μια ανανέωση του πληθυσμού και μάλιστα σε έφθετο χρόνο. Πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το σχέδιο διαχείρισης για το ευρωπαϊκό χέλη είναι καλό και θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε το στόχο μας και για τα, κράτα, για τα κράτη-μέλη που δεν έχουν σχέδιο διαχείρισης, που δεν έχουν λάβει μέτρα. Ε, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα άσκησης πίεσης ε, κατά των χωρών ε, μελών αυτών που ολιγορούν. Τι πρόκειται να γίνει, τι πρόκειται να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ δεν έχω πίστη για την αποτελεσματικότητα της πολιτικής για την ανασύσταση του πληθυσμού. Γιατί το να παίρνουμε τους γόνους από... και να τους μεταφέρουμε το ένα σημείο στο άλλο, δεν ξέρω αν είναι αποτελεσματικό. Βέβαια, εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονας, δεν έχω επιστημονικές γνώσεις για τα θέματα αυτά. Αλλά φαντάζομαι ε, εσείς θα το ξέρετε. Μήπως όμως υπάρχουν άλλα μέτρα που είναι πιο αποτελεσματικά. Όπως είπα, το θέμα είναι γνωστό και δεν είναι μόνο θέμα Λισαβονοποίησης, προσαρμογής της ηθίκης Λισαβόνας, είναι πολύ πιο σοβαρό το θέμα. Και νομίζω ότι είναι και η ώρα να λάβουμε κάποια μέτρα. Ευχαριστώ κύριο Φερέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ εκείνο από τις επιφυλάξεις και τις ανησυχίες που διατυπώθηκαν και όπως είπε και η Σαμπέλα, το απόθεμα χελιού είναι ενιαίο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, η εξέλιξή τους στους, ε, στις υδρογραφικές λεκάνες Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι διαφορετική, αλλά το απόθεμα του χελιού είναι ενιαίο. Επίσης, ε, υπάρχουν μεγάλες διακοιμάνσεις ό,τι αφορά το ποσοστό ανάπτυξης στις διάφορες ε, λεκάνες. Όσο μεγαλύτερο είναι το μήκος, το γεωγραφικό μήκος, τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό αναπαραγωγής. Ενώ στους, στα Δέλτα, υπάρχουν μεγαλύτερες εκβολές των ποταμών, έχουμε μεγαλύτερα ποστά αναπαραγωγής. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι υπάρχουν σοβαρές διακυμάνσεις μεταξύ των διαφόρων υδάτινων λεκανών που αναπτύσσονται τα χέλια και αυτές οι διακυβα... αυτέ αυτές οι διαφορές μπορούν να μας οδηγήσουν σε σημαντικές διαφορές της κατάστασης του ελευτικού αποθέματος ανάλογα με τον τόπο, το, τη γεωγραφική τοποθεσία, τα χαρακτηριστικά του, της υδρογραφικής λεκάνης, άλλο αν μιλούμε για ποτάμι, άλλο αν μιλούμε για εκβολή ποταμού ή δέλτα ποταμού. Και επαναλαμβάνω, οι διαφορές είναι τεράστιες. Και θα ήθελα και τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το, για το θέμα αυτό. Ξέρω ότι σε ό,τι αφορά πληθυσμούς ε, στο, στην Νότια Ευρώπη δεν υπάρχουν στοιχεία για να αποτιμηθεί η παρούσα κατάσταση του αποθέματος χελιού. Μερικές φορές χρησιμοποιήθηκαν τα στοιχεία για τους πληθυσμούς χελιών του Βορρά. Παρά τη διαφορά που υπάρχει, δεν μπορούμε να παίρνουμε στοιχεία του Βορρά και να κάνουμε προσωμείωση ε, γιατί επαναλαμβάνω υπάρχουν τελα, τεράστιες διαφορές της κατάστασης ε, των πληθυσμών χελιών στο βορρά και στο νότο. Δεν μπορούμε να αξιοποιούμε στοιχεία του βορρά που είναι πολύ πιο συγκεντρωμένα και ακριβή και να τα προβάλλουμε απλώς στα, στις χώρες του νότου. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε κατά πολύ τη συγκέντρωση στοιχείων και τις γνώσεις που έχουμε για το χέλι και την κατάσταση των αποθεμάτων στο νότο. Επίσης ε, γνωρίζουμε ότι πολλοί παράγοντες συμβάλλουν ε, στην ε, απειλή, αλλά δεν ξέρουμε ποιος είναι ο βαθμός της συμβολής και της επιρροής. Λαθρεμπόριο, για παράδειγμα, η παράνομη αλία των νεαρών χελιών, των μικρών χελιών. Συμβάλλει σίγουρα στην, στην απειλή, αλλά σε τι βαθμό. Επίσης, στη Νότιο Ευρώπη, στην Πορτογαλία, έχουμε σημαντικές διαφορές ε, σε ό,τι αφορά τη στάθμη των νερών των ποταμών. Η δημιουργία των φραγμάτων μερικές φορές, το φραχτό δημιουργεί πρόβλημα. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός και ίσως ε, θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη ε, την προσπάθεια μετριασμού των περιβαλλοντικών συνεπειών εξαιτίας κάποιων ε, κατασκευών φραγμάτων, για παράδειγμα, φραχτών. Έγιναν κάποιες πανεπιστημιακές προσπάθειες το τελευταίο καιρό για να μετριαστούν αυτά τα περιβαλλοντικά αποτελέσματα, αλλά δεν ευωδόθηκαν δυστυχώς. Υπάρχει κατακαιρματισμός λοιπόν των οικοσυστημάτων, των βιοτόπων, των χελιών, που συμβάλλει επίσης ε, στον περιορισμό του αποθέματος ή οι ασθένειες. Υπάρχουν μερικές ασθένειες που είναι ευρέως διαδεδομένες και δυστυχώς ε, αποδεκατίζουν τον πληθυσμό των χελιών. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες που επηρεάζουν ε, την κατάσταση του αποθέματος, αλλά υπάρχει άγνοια γενικώ και για την κατάσταση των πληθυσμών χελιών και για τη συμβολή του κάθε παράγοντα στην ε, γενικότερη απειλή κατά του αποθέματος. Και αυτό είναι που με προβληματίζει ιδιαίτερα. Γιατί δεν βλέπω καμία ελπίδα ή καμία πιθανότητα να αλλάξει η κατάσταση, δυστυχώς. Τουλάχιστον στην Πορτογαλία. Το πρόβλημα είναι πια χρόνιο. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έλλειψη στοιχείων για την αλληλευτική πολιτική. Μιλούμε για μια πολιτική που είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, μην είναι αποκλειστική ευρωπαϊκή πολιτική α, της α, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά το κόστος η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συγκέντρωση δεδομένων, για παράδειγμα, το επιρρύπτει στα κράτη-μέλη. Και δεν ξέρουμε τι κατάσταση επικρατεί σε χώρες όπως η Πορτογαλία, σε άλλες χώρες του Νότου που βρίσκονται σε προγράμματα διάσωση, Ελάχιστες δυνατότητες επιστημονικές και τεχνικές έχουμε για να αξιολογήσουμε δημόσιες πολιτικές ε, στην Αλία και δεν τις χρησιμοποιούμε ούτε καν αυτές η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που ασκεί πίστα στα κρατημέλη λέγοντας «προσοχή, δεν μας δίνετε τα στοιχεία που σας ζητάμε», αλλά η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα σχέδια παρέμβασης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απολύει δημοσίους υπαλλήλου. Ε, περικόπτει δραστικά τους, προπολογισμού τους προϋπολογισμούς των πανεπιστημίων, οπότε τη λίγη δυνατότητα εμπειρογνωμοσύνης που έχουμε πανεπιστημιακή και τεχνική την ε, φημώνουμε εξαιτίας της έλλειψης μέσων. Οι επιστήμονες αυτό είναι το πρώτο που μας λένε, ότι όλος παραδόξως τα μόνα στοιχεία που έχουν είναι στοιχεία από την αλληλεία και τις εκφορτώσεις αλληλευτικών προϊόντων και λένε μην απαγορεύσετε αυτή την γιατί το λίγο που ξέρουμε για την κατάσταση των αποθεμάτων αυτών είναι χάρη στα στοιχεία που έχουμε για την αλία. Άλλο, άλλη πηγή πληροφοριών δεν έχουμε. Εγώ δυστυχώς δεν έχω λύση για τα προβλήματα που επισήμανε η Ισαβέλα και μάλιστα προσθέτω και τα δικά μου προβλήματα, αυτά που εντοπίζω εγώ ως προβλήματα. Θα πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας μέλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φεραίρο, κύριος Γκάλεχερ. Quite brief, but my particular interest in uh, goes back some few years ago when εδώ και κάποια χρόνια στην Ιρλανδία αποφασίσαμε να σταματήσουμε την αλία, να κλείσουμε την αλία των χελιών. Μας είπαν θα χρειαστούμε 99 χρόνια πριν να αποκατασταθεί το απόθεμα. Έτσι μας είπαν τότε, αλλά φαίνεται ότι δεν ήταν ακριβής αυτή η πρόβλεψη. Ε, σε όλη την Ευρώπη γίνεται η αλληλεία. Όλοι πρέπει να παίξουμε το ρόλο μας ούτως ώστε να αποκατασταθεί το απόθεμα. Πρέπει να προστατεύσουμε τα υπάρχοντα θέλουμε να είναι βιώσιμη η αλληλεία και η προσέγγιση από τη θάλασσα των Σαργασών μέχρι την Ευρώπη. Χρειάζεται περαιτέρω έρευνα. Ίσως είναι καλή αυτή η περίοδος η χρονική που θα συζητήσουμε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αλία. Θα είναι χρήσιμο αυτό το ταμείο. Μπορούμε να διευκρινίσουμε την πλέον δεδειγμένη λύση λύση που θα προτείνουν, θα συστήσουν οι εμπειρογνώμονες. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι μειώθηκε η αλληλεία των χελιών από όταν εφαρμόστηκε πρώτη φορά ο κανονισμός που έχουμε μπροστά μας. Αναφέρομαι στα αποθέματα. Θα μπορούσαν να αποκατασταθούν τα αποθέματα στη θάλασσα των Σαργασών σε μια πιο σύντομη περίοδο στο Νότο, σε τρία χρόνια περίπου. Ε, αλλού χρειάζεται μεγαλύτερη περίοδος, 25 ε, χρόνια, στον πιο ψυχρό βορρά. Ένα νέο διαχειριστικό σχέδιο θα επέτρεπε να εφαρμόσουμε καλύτερα δράσεις ανάκτησης, αποκατάστασης, να δημιουργηθούν οι ευνοϊκότεροι όροι στην Ευρώπη. Δεν θα αναφερθώ στους λόγους για τη μείωση των αποθεμάτων, είτε αλλαγή του κλίματος, είτε είναι ρήπανση αυτή. Πιστεύω όμω ότι μια μακροπρόθεσμη λύση για να απελευθερωθούν οι μεταναστευτικές προσεγγίσεις, μεταναστευτικέ διαδρομέ. Μπορούμε να αλλάξουμε τα διάφορα φράγματα, ε, να υπάρχει προστασία στους διάφορες αντλίες, υδροελεκτρικές αντλίες κλπ. να βοηθήσουμε να περάσουν τα φράγματα όταν πηγαίνουν ενάντια στο ρεύμα. Πρέπει να κινηθούμε τώρα για να αποκατασταθεί το χέλι. Και θα πρέπει να μπουν ε, τα νέα ψάρια στους βιοτόπους που πρέπει. Είναι σημαντικός τομέας. Σωστό είναι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τώρα. και πρέπει να υποστηρίξουμε την έρευνα. Ε, και μάλιστα μέσω του Ταμείου Αλίας. Ευχαριστώ, κύριε κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. We Συνήθως ακολουθούνται διαφορετικές κατευθύνσεις. Και δεν πετυχαίνουμε εύκολα συμφωνία. Όλοι σήμερα έδειξαν ότι ανησυχούν και πολύ για το χέλι. Ίσως γιατί πνοτιζόμαστε από ένα πολύ ρομαντικό πλάσμα. Περιμένει για την Πανσέλινο. Περνά τον Ατλαντικό, πάει κόντρα στο ρεύμα, ζευγαρώνει και ξεψυχάει. και θα πρέπει να βρούμε εύκολες λύσεις όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται. Αυτή τη φορά δεν τα βρίσκουμε. Δεν βρίσκουμε τις λύσεις. Περιμένουμε να δώσει τις απαντήσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ίσως είμαστε υπερβολικά αισιόδοξοι. ρίχνουμε τον μπαλάκι στην ε, Κομισιόν. Αν δώσουν κάποια απάντηση, καλώς. Αν δεν βρουν οι, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απάντηση, θα ψάξουμε εμείς να βρούμε απάντηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ισαβέλα που μας ε, ενημέρωσε για την ε, κατάσταση. Αναμφισβήτητα πρέπει κάτι να κάνουμε. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να κινηθούμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε ή να κινηθούμε τώρα. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Θέλω να ακούσω ότι έχει να πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαι από τη Βόρεια Δανία και θυμάμαι ότι εδώ και 50 χρόνια στο Λινφιόρντ, στο βορρά της Δανίας, αλλιεύαμε πολύ το χέλι. Όλος ο κόσμος ψάρευε χέλια. Για μας το χέλι αντιπροσωπεύει πολλά πράγματα. Για το Λινφιόρντ, Σήμερα είδαμε από τη συζήτηση ότι υπάρχει μικρή πρόοδος, αλλά όχι μεγάλη. 1% μας το είπε η Σαβέλα. Έχει μειωθεί το απόθεμα 5% ε, σε όλο τον κόσμο. Σε σχέση με το απόθεμα εδώ και 50 χρόνια. Είναι 5% σήμερα στον υπόλοιπο κόσμο. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Γιάννης για το σχέδιο αποκατάστασης των αποθεμάτων στις διάφορες χώρες. Είναι ανησυχητική κατάσταση. Από ό,τι κατάλαβα, υπάρχουν εκείνοι που κινούνται για την αποκατάσταση των αποθεμάτων Έχουμε μικρότερο 5% των νέων ηχθείων. πρέπει να δούμε και το ποσοστό επιβίωσης των νέων που γίνονται για να γίνουν ενήλικα. 50% των νεογνών επιβιώνουν για να γίνουν ενήλικα ψάρια. Λένε ότι, δεν, ότι θα πρέπει να μειωθεί η αλία. Η δραστηριότητα ελευτική όμως ε, πώς θα επηρεαστεί Πώς θα αλλάξουμε τα κίνητρα που έχουν οι αλληλείς να ψαρέψουν το χέλι. Αν μια εταιρεία παραλαμβάνει 5 εκατομμύρια νέο να χρησιμοποιεί τα 2 εκατομμύρια και πουλάει τα υπόλοιπα, τι γίνεται. Δεν θα έχει δυνατότητα να κινηθεί στο μέλλον αυτή η εταιρεία. Το ερώτημα είναι, αν είναι χρήσιμες αυτές οι δραστηριότητε εάν χρησιμοποιηθούν για αποκατάσταση τοποθέματος αυτά τα νέα ψάρια, τα δύο εκατομμύρια το χρόνο. Ε, θα ήθελα να ξέρω, υπάρχουν και άλλες ε, δοκιμές που έγιναν όσον αφορά τις προσπάθειες αποκατάστασης. Χρειάζεται κάτι να κάνουμε όμως. Και τελευταία η κυρία Φράγα. Θα είμαι λακωνική. Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Λόβιν Αν δηλαδή θα πρέπει ε, να δεχτούμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για, για την επιτροπολογία και την προσαρμογή στη συνθήκη της Λισαβόνας να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Εγώ γενικώ πιστεύω θα πρέπει να περιοριζόμαστε στην προσαρμογή της επιτροπολογίας και στη διαδικασία αυτή της ε, ευθυγράμμισης με τη συνθήκη της Λισαβόνας και να μην επεσερχόμαστε σε θέματα ουσίας και σε μεταγενέστερη φάση να δούμε αν έχει νόημα να ζητήσουμε για τα ουσιαστικά θέματα πρόταση αναθεώρηση του κανονισμού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ερώτηση κυρία Λόβιν θα προτιμούσα στην περίπτωση αυτή να περιοριστούμε μόνο στην προσαρμογή της επιτροπολογίας και στην ευθυγράμμιση με τη συνθήκη της Λισαβόνας και να μην επισέρθουμε σε πιο ουσιαστικά θέματα. Αυτό μας ενδιαφέρει, να προσαρμόσουμε την επιτροπολογία. Και αν θεωρούμε ότι για ουσιαστικά θέματα ε, χρειάζεται τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού, αυτό μπορούμε να το ζητήσουμε αργότερα. Πάντως, στα πλαίσια της διαβούλευσης θα πρέπει να περιοριστούμε στο τυπικό θέμα, στην προσαρμογή της επιτροπολογίας. Δεν θα επισέλθω στην ουσία του θέματος, γιατί γι' αυτό μίλησαμε πολύ περισσότερο. Εγώ λέω, επαναλαμβάνω, να περιοριστούμε στην προσαρμογή στην επιτροπολογία. Καλώς ο κύριος Θεοφίλου τώρα για να μας παρουσιάσει τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλές ε, ερωτήσεις υπευλήσαν, πολλές παρατηρήσεις. Θα προσπαθήσω να τις ε, απαντήσω με τη σειρά και να μην παραλείψω καμία. Καταρχήν, ε, χαιρόμαστε για το ζωηρό ενδιαφέρον της κυρίας Λόβιν και την πρόταση της για την βελτίωση, την αναθεώρηση του κανονισμού. Θα ήθελα όμως ε, να διευκρινίσω ότι μιλάμε εδώ για δύο διαφορετικές διαδικασίες. Η μία προβλέπει την ευθυγράμμιση με τις Συνθήκη της Λισαβόνας, που είναι μια απλούστατη διαδικασία. Και έχουμε ξεκινήσει και τη διαδικασία της τροποποίησης της ουσίας του κανονισμού. Κάτι που προβλέπεται στον ε, ισχύοντα κανονισμό. Με βάση λοιπόν τις εκθέσεις προόδου που λάβαμε από τα κράτη-μέλη, τα τελευταίου τους τελευταίους μήνες και λαμβάνοντας υπόψη και τα επιστημονικά πορίσματα και συμβουλές, η ετήσια με επιστημονική συμβουλή της ISIS που αναφέρθηκε, αλλά και το αίτημα προς την ΆΙΣΙΣ που θα εξεταστεί από την STCF, την Επιστημονική, Τεχνική και Οικονομική Επιτροπή Ελίας, την ΕΤΟΕΑ, με βάση όλα αυτά τα στοιχεία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταρτήσει μια περιεκτική έκθεση πρόοδου και θα την υποβάλει πριν τα τέλη του τρέχοντο έτου. Θα υποβάλουμε την έκθεσή μα στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και υπό το φω αυτή της έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δύναται να προτείνει τροποποίηση του κανονισμού. Δηλαδή τροποποίηση της ουσίας, του ουσιαστικού περιεχομένου του κανονισμού όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα για τα διάφορα μέτρα, τα αλληλευτικά και μη, όλα αυτά θα αξιολογηθούν με βάση τις εκθέσεις πρόοδου που θα μας υποβάλουν τα κράτη-μέλη. Τώρα, ως προς τα σχόλια που σημείωσα εδώ, πρώτον, ο στόχος ανασύστασης του αποθέματος που τέθηκε στο 40% ο στόχος αυτός, 40% για την ανασύσταση, είναι μακροπρόθεσμος, απότερος στόχος. Ούτε οι επιστήμονες, αλλά ούτε και οι αρχές διαχείρισης, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν περιμένουν να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος ανασύστασης του 40% μέσα σε 2-3 χρόνια κατά την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης. Επαναλαμβάνω, ο στόχος αυτός είναι πιο μακροπρόθεσμος και με βάση τις επιστημονικές ε, γνωματεύσεις, στην καλύτερη περίπτωση θα υλοποιηθεί σε δύο-τρεις γενιές χελιών και αν λάβουμε υπόψη ότι μια γενιά διαρκεί από 5 με 20 χρόνια, κάντε τον απλό πολλαπλασιασμό και διαπιστώνετε ότι θα χρειαστούμε 10 με 60 χρόνια και μερικές φορές ακόμη και περισσότερο για να πετύχουμε την ανασύσταση του αποθέματος χελιού. Δεν περιμένουμε λοιπόν από τα κράτη-μέλη να υλοποιήσουν αυτό το στόχο μέσα σε 2-3 χρόνια. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις σάιτες ε, και την ταξινόμηση, ε, το Ευρωπαϊκό Χελί περιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή στο παράρτημα 2 της σάιτες, κάτι που ε, επιτρέπει την αλλιευσή του υπό όρους. Αλλά το εμπόριο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός απαγορεύεται και σε περισσότερα για να μην πω σε όλα τα σχέδια διαχείριση των κρατών μελών εξαρτάται από την εισφορά του τομέων αλλιές και δετοκαλλιέργειας που είναι αλληλένδετη και από αυτούς εξαρτάται η υλοποίηση του στόχου. Δηλαδή, ε, αν δέχτηκε ο ψαράς να αφήσει μερικά από τα χέρια που αλλιεύει. Οπότε, αν αναβαθμιστεί το χέλι και περάσει από το παράρτημα 2 στο παράρτημα 1 του ΣΑΙΤΕΣ, θα απαγορευτεί και η έλλειψη, όχι μόνο η εμπορία. Κάτι που σημαίνει κατάρρευση των σχεδίων διαχείριση των κρατών μελών για το χέλι. Πολλές ερωτήσεις ε, υπευλήσαν από τον κύριο Νίλσον. Ποια είναι η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για τα υφιστάμενα σχέδια διαχείρισης διαπιστώνουμε ότι κάποιες χώρες κάνουν πολύ μεγαλύτερη πρόοδο από άλλες. Και αυτό για πολλούς και διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, λόγω της γεωγραφικής κατάστασης, της βιολογικής κατάστασης, αλλά και της κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης ε, που διαφέρει από χώρα σε χώρα και από λεκάνη σε λεκάνη, από ποτάμι σε ποτάμι. Σε μερικές φορές έχουμε έντονη αλήψη, σε άλλες όχι. Ε, ορισμένα ποτάμια ε, είναι μπλοκαρισμένα και από οικονομική άποψη ήταν αδύνατο να αρθούν τέτοια κολλήματα, ενώ σε άλλε περιπτώσει, σε άλλα ποτάμια, έχουμε απόλυτη ελευθερία, κανένα μπλοκάρισμα. Γι' αυτό και αφήσαμε στι χώρε να επιλέξουν τα καταλληλότερα μέτρα, λαμβάνοντα υπόψη τι ιδιομορφίε του για να πετύχουν το στόχο ανα, ανασύσταση. Δεν θέλαμε να υποχρεώσουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν όλα τα, να εφαρμόσουν τα, τα ίδια μέτρα ε, για να υλοποιήσει το στόχο ανασύσταση στα ποτάμια τους. Τώρα, ω προ τη δεύτερη ερώτηση. Επαναλαμβάνω, ο στόχο τη ανασύσταση είναι μακροπρόθεσμος. Η ανασύσταση θα πετήσει δεκαετίες, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Τώρα, τι γίνεται με τα κράτη-μέλη που δεν συμμορφώνονται. Μερικές χώρες δεν υπέβαλαν ακόμη σχέδια διαχείρισης όπως θα όφυλαν και όπως προβλέπεται στον κανονισμό. Σε τέτοια περίπτωση ίσως σου επιβληθεί υποχρεωτική μείωση 50% της αλίας χελιού. Τώρα, ανασύσταση η ανανέωση του πληθυσμού αναφέρθηκε από πολλούς είναι ή ο τεχνητός εμπλουτισμός αμφιλεγόμενη πρακτική από επιστημονική άποψη η ο τεχνητος εμπλουτισμος αμφιλεγομενη πρακτικη απο επιστημονικη αποψη η ISIS μας λέει ότι ίσως το restocking δεν συμβάλλει όσο θα επιθυμούσαμε. Ταυτόχρονα η ISIS αναγνωρίζει ότι αν το restocking, αυτός ο τεχνητός εμπλουτισμός, γίνει με τους σωστούς όρους, με σωστό χρονισμό και στη σωστή τοποθεσία, ίσως συμβάλλει στην υλοποίηση του στόχου ανασύστασης. Το restocking πάντως είναι μια μέθοδος που θα εξεταστεί στη συζήτηση στα πλαίσια της ουσιαστικής τροποποίησης του κανονισμού. Σε ό,τι αφορά την επιστημονική γνώση μέσω των σχεδίων διαχείρισης και μέσω των παράλληλων προγραμμάτων. Έχουμε βελτιώσει λοιπόν την επιστημονική μας γνώση και θα συνεχιστεί αυτή η βελτίωση, κάτι που θα επηρεάσει τα μέτρα διαχείρισης που θα προτείνουμε σε αρχές του επόμενου έτους. Αυτό είναι ένα δεικτικό χρονοδιάγραμμα και πρόβλεψη. Τώρα, για πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, σε ό,τι αφορά τις επιστημονικές γνωματεύσεις, περιμένουμε την γνώμη της ISIS ε, στα μέσα Ιουνίου και όπως και απαιτεί ο κανονισμός ε, για το χέλι. Η ΕΤΟΕΑ θα τροποποιήσει τα μέσα Ιουλίου την γνωμάτευση αυτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη όλα αυτά τα, όλες αυτές τις προτάσεις στην τροποποίηση του κανονισμού που θα υποβάλει σε αρχές του 2014. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Θεοφίλου, κυρία Λέβιν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους ε, που συμμετείχαν σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Τους ευχαριστώ όλους. Έχω κάποια σχόλια. Θα ήθελα να πω στον κύριο Κιούν. ανησυχείτε πολύ για την έλλειψη δεδομένων κτλ. Ναι, προφανώς υπάρχουν τεράστια κενά στην ενημέρωση σε ό,τι αφορά το πού αναπαράγονται τα χέλια, ποιε είναι οι αιτίε της ε, μείωση, τη επιδείνωση του αποθέματο, αλλά υπάρχουν πολλά δεδομένα, πολλά στοιχεία για το τι γίνεται με την ε, μετανάστευση και την, ε, ε, των μικρών χελιών προς την Ευρώπη και την διαφυγή των συμμόχελων. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να δείτε και τα στοιχεία αυτά και τις συστάσεις της ΆΙΣΕΣ, γιατί και εκεί υπάρχουν πολλές αναφορές στους λόγους για τους οποίους μειώθηκε το απόθεμα. Για τον κύριο Φερέιρα, πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλιά σας. Μιλήσατε για ένα, ότι όντω είναι ένα το απόθεμα, αλλά είπατε ότι μπορεί να είναι διαφορετικοί πληθυσμοί. Δεν υπάρχουν διαφορετικοί πληθυσμοί. Ένα είναι το απόθεμα, ακόμα και αν υπάρχει ε, υπάρχουν περισσότερα αποθέματα σε κάποιες ε, λεκάνες του ενός ή του άλλου είδους χελιού. Παρ' όλα αυτά το συνολικό απόθεμα βρίσκεται σε ε, πολύ ε, δυσμενή κατάσταση. Τώρα, για τα, για τα εμπόδια που υπάρχουν για τους ε, ε, διάβλους μετανάστευσης. Αν δείτε την ε, αναφορά της ISIS και το πότε ξεκίνησε αυτή η μεγάλη μείωση, ήταν τη δεκαετία του 80. Δημιουργήσαμε πολλά υδροελεκτρικά εργοστάσια εμείς ήδη από πολύ πιο πριν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εν πάση περιπτώσει, υπήρξε τεράστια εκμετάλλευση των ποταμών. Ήδη εδώ και 100 ή και 50 χρόνια. Σίγουρα δεν άρχισε το κακό πριν από 20 χρόνια. Γι' αυτό και οι επιστήμονες λένε ότι υπάρχει και η πίεση της υπεραλίευσης, που είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την επιδείνωση. Τώρα, για το κόστος της εφαρμογής. Συμφωνώ. Η Ευρώπη όντως βρίσκεται υπό οικονομική κρίση, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για το γιατί τα κράτη-μέλη ήδη από πιο πριν που δεν υπήρχε οικονομική κρίση δεν έκαναν τίποτα και γιατί έχουν υπάρξει αυτές οι τεράστιες καθυστερήσεις ε, στην υποβολή ε, των, σχεδίων διαχείρισης των κρατών μελών πραγματικά τα κράτη-μέλη τα έχουν πάει χάλια σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν νομίζω ότι φταίει η οικονομική κρίση γι' αυτό. Εδώ και 10-15 χρόνια τα κράτη-μέλη δεν τα πάνε καλά. Ο μόνος τρόπος για να αποκτήσει κανείς ε, δεδομένα είναι η αλία. Και αυτό το επιχείρημα με κάνει να θυμάμαι πάντα τους ε, Ιάπωνες και τους Ισλανδούς όταν ε, λένε ότι πρέπει να αλλιεύουν φάλαινες για να έχουν τα δεδομένα. Ε, εντάξει, αυτό δεν είναι σοβαρό επιχείρημα. Δεν μπορούμε να αλλιεύουμε μόνο για, μόνο να, για να μετρούμε πόσα αλλιεύματα έχουμε και πόσο μειώνονται τα αποθέματα χελιού. Αυτό δεν βγάζει νόημα. Νομίζω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε κονδύλια για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε ναι, για να αλλιεύσουμε ίσως τα χέλια και μετά να τα απελευθερώσουμε. Έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη εδώ από τη Σουηδία που κάνει έναν υπολογισμό για το ποιο είναι το κόστος της διαχείρισης του χελιού στην Σουηδία. Μιλούμε για την έρευνα, μιλούμε για την ανασύσταση του αποθέματος, για όλα τα διοικητικά, για τους ελέγχους, για όλα και φτάνει στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Η αξία της αλληλείας χελιού στην Σουηδία είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε πληρώνουμε περισσότερο για τη διαχείριση παρά για την αλίευση. Υπάρχει λοιπόν, υπάρχουν κονδύλια. Το θέμα είναι πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Και νομίζω ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε ώστε να ε, μπορέσουμε να αλλιεύσουμε χέλια από περιοχές όπου μπορούν να γίνουν ε, μεταφορές σε άλλες περιοχές και να μπορούν να επιβεώσουν. Κύριε Γκάλαγκερ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Χρειάζεται ένα ενιαίο σχέδιο διαχείρισης για την Ευρώπη. Αυτό πραγματικά ήταν ένα τεράστιο εγχείρημα, πείραμα, του, που αποδεικνύει πως τα κράτη-μέλη δεν έκαναν τη δουλειά τους σε ό,τι αφορά την περιφερειοποίηση. Στην κοινή, αγροτική, στην κοινή αλευτική πολιτική τα κράτη-μέλη έχουν πολλή ελευθερία και τελικά δεν κάνουν ό,τι πρέπει. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ώστε να υπάρχει μία συγκρίσιμη μέθοδος για όλα τα κράτη-μέλη. Κύριε Κρίστανσεν, μιλήσατε για την ανασύσταση του αποθέματος. Ίσως να έπρεπε να πω δύο πράγματα παραπάνω για το γιατί η ISIS δεν ε, υποστηρίζει αυτό το επιχείρημα. Καταρχάς, το ανασυσταθέν απόθεμα μπορεί να καταλήξει και πάλι στην ε, περιοχή αναπαραγωγής. Γιατί αν πάρετε ας πούμε από το βυσκαϊκό κόλπο κάποια χέλια, τα, πάρετε, τα σταφίστε στην Σκανδιναβία, τα απελευθερώστε στην ε, Βαλτική θάλασσα, δεν υπάρχει καμία υποστημονική ε, απόδειξη που να λέει ότι αυτό το χέλι που έφτασε τελικά στη Βαλτική θα ξαναβρει τον δρόμο του για να φτάσει πίσω στο βυσκαϊκό κόλπο. Ίσως ε, για τον Ατλαντικό να μπορούν να ξαναβρούν τον, ε, το δρόμο τους, αλλά αν, αν, ε, μεταφέρουμε τα χέρια σε τελείω διαφορετικά μέρη, μπορεί να μην μπορούν να βρουν πάλι το δρόμο τους πίσω. Και υπάρχουν κάποιες μη δημοσιευμένες μελέτες που λένε ότι κάποιο ανασταθέν από, απόθεμα κατάφερε να φτάσει πίσω, από πίσω στη Σκοτία από τη Σκανδιναβία. Αλλά αυτό δεν είναι ο κανόνας. Οπότε ίσω να πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και την ε, ρήτρα προφύλαξη ω προ αυτό. Μετά υπήρξε ένα ερώτημα για το πόσα μικρά χέλια επιβιώνουν αν τα πάρετε και τα πάτε από τη μία περιοχή στην άλλη. Μήπως μεταφέρουν ζωονόσους όταν τα μεταφέρουμε στην άλλη περιοχή. Εγώ συναντήθηκα με μία ομάδα που λέγεται η ομάδα του βιώσιμου χελιού και μου έδειξαν μία μελέτη που έκαναν για την μεταφορά και την ανασύσταση ε, του χελιού και κατά πόσο αυτό βοηθάει τον ευρωπαϊκό πληθυσμό χελιού. Και σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη μελέτη, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι μπορεί όντως να συμβάλλει στην ανασύσταση, στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού αποθέματος. Αλλά στη σελίδα τρία της περίληψης, ο συγγραφέας της έκθεσης λέει ότι δεν μπορούμε να πούμε κατά πόσο αυτό σημαίνει συνολική αύξηση σε σύγκριση με το να αφήσουμε τους γόνους εκεί που είναι. Αν αφήσετε δηλαδή τους γόνους εκεί που βρίσκονται, δεν θα πεθάνουν κατά τη διάρκεια της αλίευσης, δεν θα πεθάνουν κατά τη διάρκεια της ε, μεταφοράς, δεν υπάρχουν ερωτηματικά για το κατά πόσο θα μπορέσουν να φτάσουν πίσω στη θάλασσα των σαργασών κτλ. Αυτό λέει η έκθεση. Είναι δηλαδή ο κλάδος που την ε, ε συνέταξε αυτή την έκθεση. Λαμβάνοντα υπόψη και τι ε, προτάσει τη που είναι πάντα πολύ συντηρητική στα σχολεία τη ό,τι αφορά τι μεταφορέ των χελιών. Ε, πρέπει λοιπόν να το δούμε. Και επίση η ΆΙΣΕΣ λέει ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει επιπλέον ε, γόνος στην Ευρώπη ώστε να μπορεί να ανασυσταθεί ή να μεταφερθεί. Οπότε για, την, για τα όσα μας είπε η Κομισιόν τώρα. Καταλαβαίνω ότι ο στόχος είναι μακροπρόθεσμα να φτάσουμε το 40% και όχι για τα 2-3 χρόνια που μιλούμε. Εντάξει, ως εδώ. Αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν και με το πόσο αόριστα είναι τελικά τα πράγματα. Υπάρχουν παντού κενά είναι μακροπρόθεσμο. Ε, μιλούμε για δυο τρει γενιέ χελιών, ε, που ε, μια γενιά μπορεί να είναι 5 με 20 χρόνια, δηλαδή μιλούμε για 10 με 60 χρόνια διάρκεια. Οπότε... Πρέπει να, να τα ορίσουμε λίγο πιο καλά αυτά για το τι σημαίνει διαφυγή, ποιο, για ποιο κύκλο ζωής μιλούμε. Είναι τόσο αφηρημένα που είναι αδύνατο για οποιοδήποτε να ελέγξει αν όντω τα κρατημέλη τηρούν τα προγράμματα ή όχι δεν, δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλή αυτή η προσέγγιση. Είπατε βέβαια ότι αν εφαρμόσουμε το παράρτημα 1 της ΣΑΙΤΕΣ, τότε όλα τα ε, προγράμματα διαχείρισης θα κατέρεαν. Ναι, αυτό αληθεύει. Πέραν, ε, εκτός από την Ιρλανδία, γιατί η Ιρλανδία υπέβαλε ένα σχέδιο και δεν έχει αλλιεύσει χελιού πια. Οπότε είναι δυνατό να υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης χελιού που δεν θα περιλαμβάνει αλία χελιού. Και επίσης ε, μιλήσατε για την όλη διαδικασία, την εξηγήσατε. Εγώ έθεσα το ερώτημα στην Κομισιόν το Μάιο του 2011 και η Επίτροπος Δαμανάκη απάντησε ότι δεν μπορεί να εξαιρεθεί ότι τα ε, επίγοντα μέτρα που προτείνονται από την Κομισιόν για την αντιμετώπιση των σοβαρών ανησυχιών που υπάρχουν και οι ανησυχίε αυτές ήταν τα μέτρα της, ε, ότι τα μέτρα ανασύστασης δεν είναι ε, επαρκή. Ε, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να ρωτήσω και πάλι την Κομισιόν. Η Κομισιόν δεν προβλέπει να εφαρμόσει, να αναλάβει μάλλον έκτακτα μέτρα όσο τροποποιεί το πρόγραμμα και όσο περιμένει τις, εκτι, τις εκτιμήσεις της ISIS και της ΤΕΚ. Αυτά, Πρόεδρε, από μένα και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Muy bien, pues. Ευχαριστώ. Θέλει άλλος κανείς το λόγο? Όχι. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημέρης διάταξης που είναι το 7, αυτό που αναβάλαμε από χθε. Έθεσα μια σύντομη ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μήπω μπορούσατε να της δώσετε το λόγο. Ε, δεν ε, κάνατε νόημα κύριε θεοφιλο; Γι' αυτό δεν σας έδωσα το λόγο. Φυσικά, σας ακούμε. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προφανώς δεν μπορώ να αποφασίσω προσωπικά τώρα. Πρέπει να επαναλάβω την ίδια απάντηση ότι είναι κάτι εφικτό. Κατεπήγοντα μέτρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Από ό,τι γνωρίζω όμως, δεν σχεδιάζουμε τώρα κάτι τέτοιο. Δεν είναι αδύνατον πριν την ε, τροποποίηση, αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να κάνουμε κάτι τέτοιο τώρα. Ωραία. Τότε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 7 και ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Νικολέσκο που είχε την καλοσύνη χθε να δεχτεί αναβολή του σημείου του για σήμερα. Αφορά την τροποποίηση του κανονισμού 850 του 98 για τη διατήρηση των αλληλευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασία των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών. Ήδη το Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας παρουσίασε την ε, πρότασή της και σήμερα θα έχουμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων εισηγητής μας είναι ο κύριος Νικολέσκο, παραλαμβάνω, στον οποίο και δίνω το λόγο αμέσω. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομο. Έχουμε μια έκθεση που αφορά τι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια έκθεση που δεν δημιουργεί μεγάλα προβλήματα. Όμω έχουμε δύο θέματα τα οποία αφορούν την διατήρηση των αληφτικών πόρων, την έκθεση Γκάλαγκερ η οποία ήδη ψηφίστηκε και αυτή την έκθεση. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα δύο θέματα εξετάστηκαν ξεχωριστά. Στην πρόταση ευθυγράμμιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμπερίλαβε τροποποίησει για τα άρθρα 4-4Γ, 7,8, 8-4 κλπ. Ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο. Άλλο πρόβλημα, για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να ανασταλούν εκτελεστικές πράξεις για τα στοιχεία που αφορούν την ευτική προσπάθεια, αλλά μόνο για τα ύδατα Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου προτείνει συγκεκριμένα μέτρα. Υπάρχουν και άλλες προ διευθέτηση λεπτομέρειες. Θέλω τις παρατηρήσεις όμως των συναδέλφων για να ετοιμάσω το κείμενο του σχεδίου εκθέσεώς μου. Ευχαριστώ. Καλώς θέλει. Κανείς το λόγο. Κυρία Φράγκα. Δύο σχόλια έχω. Ο κανονισμός αυτός ε, και η προσαρμογή της επιτροπολογίας ε, στον κανονισμό τεχνικών μέτρων δεν θα έχει πια νόημα από τη στιγμή που τεθεί σε εφαρμογή μεταρρύθμιση τη κοινή αλληλευτικής πολιτική. Γιατί θα κληθεί αμέσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει τι κατάλληλε προτάσει για να αντικαταστήσει το συγκεκριμένο κανονισμό. Βέβαια, στο μεταξύ πρέπει να κάνουμε την προσαρμογή της επιτροπολογίας. Πάντως ο κανονισμός αυτός ε, είναι καταδικασμένος να εξαφανιστεί σχετικά σύντομα. Και επιτρέπω, επαναλαμβάνω συγγνώμη αυτό που είπα χθε ε, για την απεριόριστη εκχώρηση ε, εξουσιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις κατεξουδότητες πράξεις. Εγώ προτιμώ να υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός και αυτό που συστηματικά εγκρίνουμε είναι η τριετία. Ούτως ή άλλως ε, πριν την τριετία θα καταργηθεί αυτός ο κανονισμός. Αλλά εν ώψη το... δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακριβώς με τη μεταρρύθμιση ΚΑΠΑΣ, Θέσουμε και καταληκτικό χρονικό όριο για τον κανονισμό αυτό και τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Θέλει το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να απαντήσω σε αυτά που είπε ο κύριος Νικολέσκου για το άθρο 34, παράγραφος 6. προσπαθούμε να άρουμε μέτρα για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Αφορά συγκεκριμένα μέτρα και τη ζώνη των 12 μιλίων ε, όσον αφορά την αλία και αφορά τα σκάφη του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. Δεν είναι νέος κανόνας. Συμπεριλαμβανόταν ήδη στο άρθρο. Ευθυγραμμίζουμε αυτό το άρθρο με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Ευθυγραμμίζεται και που δεν είναι αντιμετωπίζονται διαφορετικά οι διάφορες χώρες. Σε αυτά που είπε η κυρία Φράγα, απόλυτο δίκαιο έχει. Πρόθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να απαλλαγούμε από αυτό τον ε, κανονισμό. Το 50 θέλουμε με την πάροδο του χρόνου αυτό να γίνει. Ο κανόνας για τα τρία χρόνια μας βρίσκει συμφώνους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριος Νικολέσκου, δεν θέλει άλλο το λόγο. Ολοκληρώνουμε το σημείο αυτό και εξαντλήσαμε την πρωινή μας σε διάταξη. Διακόπτουμε λοιπόν και θα τα ξαναπούμε στις 3 παρουσία του Ιρλανδού Υπουργού. Γεια σας προς το παρόν.